Καλησπέρα σας ε, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι. Ευχαριστώ θερμά όσους είναι παρόντες και να τους δώσω και λίγα δευτερόλεπτα για να φορέσουν τα ακουστικά τους. Θα ξεκινήσω με τα πορτογαλικά, αλλά θα περάσω τα αγγλικά διαβάζοντας τα σημειώματα που έχει προετοιμάσει η γραμματεία. Ξεκινάμε λοιπόν όσοι ήθιστε, με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Υπάρχουν μήπως παρατηρήσεις, προτάσεις ή ενστάσεις. Όχι, οπότε εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Έγκριση των πρακτικών τώρα της προηγούμενης συνεδρίασης της 12 η Νοεμβρίου του 2012. Εγκρίνονται και αυτά και περνάμε στις ε, ανακοινώσεις του Προέδρου. Υπάρχει απευθείας αναμετάδοση της ε, Συνεδρίασή μας στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η συνεδρίαση των συντονιστών που έχει προλευθεί σήμερα ε, για τις 5.30 με 6.30 ακυρώνεται. Αν υπάρχουν κατεπήγοντα θέματα για τους συντονιστές που θα δικαιολογούσαν να επαναφέρουμε την συνεδρίαση των συντονιστών, θα πρέπει να τα δηλώσετε στον πρόεδρο ή στη γραμματεία. Πάντως, οι πολιτικές ομάδες συμφώνησαν να κυρωθεί η στη γραμματεια παντω οι πολιτικε ομαδε συμφωνησαν να κυρωθει η συνεδριαση των συντονιστών. Αν έχετε προτάσει προ τη γραμματεία για θέματα που θα πρέπει να αποφασίσουν οι συντονιστές, στείλτε σα παρακαλώ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη γραμματεία. Τώρα, αναφορά τη αποστολή μα που έγινε στις 28 με 31 Οκτωβρίου στην Ιταλία έκθεση της αποστολής αυτής που έγινε πριν από ένα μήνα περίπου. Ήδη η Γραμματεία έχει ετοιμάσει ε, την έκθεση από την αποστολή αυτή. Έχουμε, σας έχουμε στείλει μάλιστα το έγγραφο και θα ήθελα να διαβάσω το σημείωμα που έχει ετοιμάσει η Γραμματεία. Θα το διαβάσω στα αγγλικά και μετά την ανάγνωση του σημειώματος της Γραμματείας, αν κάποιος που ήταν παρόν στην αποστολή αυτή της αντιπροσωπείας στην Ιταλία από τους Αλφάμα, Γιακολίνο, Γαργάνη, Γιαννάκου, Ταπαρέλο, Μπορσελίνο, Γιώταβα, Σάσολη, Βάνα, Σις, Σμίτη, Μποργέτζο, κάποιος από αυτούς αν είναι παρόν και θέλει το λόγο μετά την ε, ανάγνωση του σημειώματος της γραμματείας πολύ ευχαρίστω για να μα παρουσιάσει τι δικέ του εντυπωσει για το τι συνέβη στην αποστολή εκείνη. Εγώ θα διαβάσω το σημείωμα τη γραμματείας στα αγγλικά. You know, Όπως ξέρετε αγαπητοί συνάδελφοι, η αποστολή τη Επιτροπή μα έλαβε χώρα στο Μιλάνο ε, Παλέρμο και Ρώμη 28 με 31 Οκτωβρίου. Ξεκινήσαμε την αποστολή στο Μιλάνο στις 29 Οκτωβρίου στο γραφείο του Κοινοβουλίου και μάλιστα εκεί είχαμε ε, συναντήσει με εισαγγελείς ε, και δικαστές από δικαστήρια της Βορείου Ιταλίας και από την αστυνομία εκπροσώπους και στις 30 Οκτωβρίου του 2012 η αποστολή της ΚΡΙΜ ξεκίνησε τις, ε, ε στην συνεδρίασή της στο εφετείο του Παλέρμο με εκπροσώπους των γραφείων καπάταξης της μαφίας και των εισαγγελέων που έδωσαν, παρουσίασαν τη θέση τους για την καταπολέμηση του εγκλήματος. Συνεχίσαμε τη συνεδρίαση στη Ρώμη στις 30 Οκτωβρίου 2012. Εκεί ακούσαμε και πάλι εκπροσώπους της αστυνομία και των ποινικών δικαστηρίων καθώς και εκπροσώπους αναθεσμικών οργάνων και επιχειρηματίες. Και μάλιστα η δική μας, η, η δική μας επιτροπή συναντήθηκε και στη Ρώμη σε διευρυμένο προεδρείο με μέλη του Ιταλικού Κοινοβουλίου από την Επιτροπή κατά της Μαφίας. Έγινε ανταλλαγή απόψεων με τους ενδιαφερομένους και ζήτησε το λόγο η κυρία Βάιλερ. Παρακαλώ, σας ακούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με τα καλά νέα. Η ε, αποστολή αυτή ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα γιατί τόσο εγώ όσο και άλλοι δεν γνωρίζαμε πόσο ε, έχει εξελιχθεί η, η Ιταλική νομοθεσία και πόσο αποτελεσματικά εργάζονται οι αρχές ε, που ε, ασχολούνται με την καταπολέμηση της ε, μαφίας. Αυτό δεν το έχω δει πουθενά ενδεχομένως. Ε, αυτό βεβαίως να οφείλεται και λόγω του ότι υπάρχει μια προϊστορία με την μαφία. Πάντως σε νομοθετικό επίπεδο η Ιταλία πρέπει να πω ότι έχει τα αποτελεσματικότερα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά, το οργανωμένο έγκλημα ε, πάντα προχωρά ένα βήμα πιο μπροστά και γι' αυτό δύο πράγματα διαπιστώσαμε που μας ανησυχούν. Αφενός, ε, λόγω της ε, χρηματοπιστωτικής κρίσης, η μαφία έχει αποκτήσει νέους πόρους για να πτήσει τις δραστηριότητες στο Νότο, αγοράζει οικόπεδα από τους ε, αγρότες, ε, αγοράζει αυτή την γη η μαφία και κατόπιν στρέφεται προς τα διευθυντικά ταμεία για επιδοτήσεις. Αυτό μέχρι εκεί ίσως να μην είναι παράνομο. Όμως ε, η μαφία είναι επαγγελματικά οργανωμένη συμμορία και για αυτό το λόγο έχει και τελείως διαφορετικές δυνατότητες να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες που υπάρχουν. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η μαφία έχει αρχίσει να μετακινείται και προς το βορρά και ε, αναπτύσσει δραστηριότητε σε τομείς που παλαιότερα δεν τους έδινε ιδιαίτερη σημασία. Δηλαδή, κατά κάποιον τρόπο έχει αρχίσει να δυσδύει σε διαρθρωτικά προγράμματα. Ακούσαμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει σχεδόν κανένα μεγάλο διαρθρωτικό πρόγραμμα, είτε πρόκειται για κανάλια, είτε για δρόμους, είτε για γέφυρες, όπου να μην συμμετέχει και η μαφία. Αυτό δεν συνέβαινε απαραίτητα κατά το παρελθόν. Τώρα είναι φαινόμενο των καιρών. Άρα δηλαδή εδώ πρέπει να επιληφθούν οι Ιταλικές αρχές αλλά και οι Ευρωπαϊκές για να δουν ε, τι τελικά συμβαίνει με τα διαρθρωτικά κονδύλια. Εγώ είδα στην έκθεσή μου ότι εκεί αναφέρεται το οργανωμένο έγκλημα δεν μπορεί να αποκτήσει τόσο εύκολα πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταμεία. Βεβαίως, ε, ε, λόγω της οικονομικής κρίσης, ε, επειδή υπάρχει έλλειψη ρευστών, πράγμα που διαθέτει η μαφία, για το λόγο αυτό μπορεί πλέον ε, να αγοράσει εκτάσεις ε, και να μπει και σε αυτά τα προγράμματα. Αυτό δημιουργεί προβλήματα. Πολύ ενδιαφέρον λοιπόν το ταξίδι. Οι υπάλληλοι του οποίου ε, συναντήσαμε ήταν ιδιαίτερα καταρτισμένοι και αυτό με εντυπωσίασε πάρα πολύ όπως και ο ζήλος με τον οποίο εργάζονται. Και αυτό θα ήταν καλό να συμβεί και σε άλλες χώρες Πολλοί λοιπόν επέκριναν ότι άλλες χώρες, η Γερμανία, η Αυστρία και άλλες ε, γειτονικές χώρες δεν έχουν τόσο διευρυμένες αρμοδιότητες και γι' αυτό δεν προχωράει η δίωξη του εγκλήματος. Αυτό λοιπόν είναι το δίλημα της Ευρώπης. Έχουμε 27 διαφορετικές ε, νομοθεσίες. Ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχουμε προχωρήσει ιδιαίτερα. Στην Ιταλία λοιπόν όλοι οι εμπειρογνώμονες ε, θεωρούν ότι πρέπει να συνεχίσουμε τις ε, προσπάθειές μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο να θεσπίσουμε τον θεσμό του εισαγγελέα ή κάτι το παρεμφερές έτσι ώστε και οι Ιταλοί να μπορούν να εργάζονται αποτελεσματικότερα. Όσον αφορά τώρα την οργάνωση του ταξιδιού αυτό το είπαν όλοι, δεν το λέω μόνο εγώ. Κοιτάξτε, δεν είναι ιδιαίτερα ε, σωστό να συναντάμε 25 υπαλλήλου σε ένα πρωινό, ε, να είχαμε λίγο περισσότερο χρόνο. Ε, την επόμενη φορά να είναι λίγο πιο βραδύς ο ρυθμός. Αλλά κατά τα άλλα πάρα πολύ ενδιαφέρον το ταξίδι. Σας ευχαριστούμε κυρία Βάιλερ. Πολύ κατατοπιστική αυτή η περιληπτική παρουσίαση της αποστολής στην Ιταλία. Δεν ξέρω αν κανείς άλλος θέλει το λόγο. Ο κύριος Νιουτοντάν, παρακαλώ. Εγώ δεν συμμετείχα σε αυτή την αποστολή, οπότε μία ερώτηση θα θέλω να κάνω, αλλά κοιτάω γύρω μου και δεν βλέπω κανέναν Ιταλό. Ή μήπως κάνω λάθος. Όχι. Μήπως τελικά ήταν ε, μια διαφήμιση για τους Ιταλούς αυτό το ταξίδι σε τρεις πόλεις ε, και ήταν καταπληκτική αυτή η διοργάνωση, ήταν περίτη υπερβολική αυτή η σπουδή ε, να συναντήσουμε τόσο πολύ κόσμο, να ταξιδεύσουμε τόσο πολύ μέσα σε λίγο χρόνο. Μήπως έτσι καταλάβαμε καλύτερα τι συνέβαινε ή το αντίθετο αποτέλεσμα είχε τελικά αυτή η αποστολή με τέτοια με Ναι και εγώ βρήκα ότι το πρόγραμμα ήταν κάπως αγχωτικό. Το Μιλάνο, γιατί το Μιλάνο, τη Ρώμη και το Παλέρνο το δυόμιση, θα είχαμε δυόμιση μέρες. Αλλά πραγματικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ιδιαίτερως προσεκτικά και μου απέφθηναν ε, πολλές ε, ερωτήσεις που αξιοποιήθηκαν όχι μόνο από τους Ιταλούς ε, συναδέλφους όπως θα το κάναμε και εμείς εδώ αλλά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πραγματικά χρησιμοποιούν αυτό το θέμα γιατί το βασικό θέμα, η διαφθορά, η απάτη είναι το πιο σημαντικό θέμα στην Ιταλία και πραγματικά θα ήθελα να υπάρξει και μεγαλύτερη δημοσιότητα και στη Γερμανία θα μου άρεσε όταν για παράδειγμα ακούμε πως το Wiesbaden που είναι η πρωτεύουσα του δικού μου κρατηδίου τι ακριβώς λέγεται και τελικά γίνεται η προσπάθεια μιας συγκάλυψης και τα πράγματα δεν βλέπουν ποτέ το φως της δημοσιότητας, θεωρώ ότι θα ήταν καλύτερο να είναι τα πράγματα όπως στην Ιταλία που όλοι ενδιαφέρονται για αυτά τα θέματα διαφθοράς. Στη Ρώμη ε, μιλήσαμε και με τους εθνικούς ε, βουλευτές που συμμετέχουν στην ε, Επιτροπή Διαφθοράς κατά της Μαφίας, στην οποία εκπροσωπούνται όλες οι πολιτικές ομάδες. Και αυτό πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέρον επίσης και ήταν όλοι παρόντες και ήταν ένα απόγευμα όπου δεν θα χρειαζόταν, ε, δεν ήταν απαραίτητο μάλλον να είναι παρόντε όλοι, αλλά είναι ένα καυτό θέμα, θέμα ύψη τη προτεραιότητα στην Ιταλία. Και ω εκ τούτου θεωρώ ότι δεν, είναι, ήταν μόνο σπατάλη χρόνου. Ε, Σοντεργάρτ. Ε, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ δεν συμμετείχα Και αυτό σχετίζεται με το γεγονό ότι είμαστε μια κάπως μικρότερη επιτροπή. Ε, αλλά είχα ε, συμμετάσχει σε ένα παρόμοιο ταξίδι στην Ιταλία με την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού και πραγματικά με κατέπληξε ο ρυθμός των ε, οργάνων που ασχολούνται με την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και της διαφθοράς. Και ε, δεχομένω θα μπορούσε ίσως να σημαίνει την εντύπωση ότι είναι υπερβολικός αυτός ο αριθμός των θεσμικών οργάνων που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Ε, γιατί ε, οι πολλοί μάγειροι όπου λαλούν πολλοί κοκόροι αργεί να ξημερώσει. Και δεν είναι δυνατό να γίνει ούτε καν ένα μεγάλο ε, έργο οικοδομικό στο οποίο να μην συμμετέχει η μαφία. Και βεβαίως ε, θα το θέμα του τι πήγε στραβά σε αυτή την αντιπροσωπεία. Δεν ε, αρκεί να υπάρχουν πάρα πολλοί αξιωματούχοι υπάλληλοι οι οποίοι να καταπολεμούν τη μαφία ή να προσπαθούν να καταπολεμήσουν την αμαθία όταν το αποτέλεσμα είναι σε κάθε κατασκευαστικό έργο τελικά να υπάρχει δίθυση συμμετοχή της ε, μαφίας. Το ερώτημα το οποίο τίθεται εδώ είναι τι πάει στραβά, τι πηγαίνει στραβά ε, εδώ. Δεν είναι ζήτημα προσώπων. Και ίσως θα μπορούσε η να προσπαθουν να καταπολεμησουν την μαφια οταν το αποτελεσμα ειναι σε καθε κατασκευαστικο εργο τελικα να υπαρχει διθυση συμμετοχη της μαφιας το ερωτημα το οποιο τιθεται εδω ειναι τι παει στραβα τι πηγαινει στραβα εδω δεν ειναι ζητημα προσωπων και ισως θα μπορουσε η αντιπροσωπεια να μας δώσει κάποιες απαντήσεις σχετικά. Τι πήγε στραβά στη, στην Ιταλία για να, μην, να προσπαθήσουν να το αποφύγουν πριν ξαναδώσω το λόγο στην κυρία Βάιλερ, να ακούσουμε και την ερώτηση τη κυρία Ματιέ, για να απαντήσετε μαζί και στις δύο ερωτήσει, κυρία Βάιλερ. Κυρία Ματιέ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ούτε κι εγώ έλαβα μέρος στην αποστολή αυτή στην Ιταλία. Λόγω έλλειψης θέσεων, γιατί όλοι ενδιαφέρθηκαν να μεταβούν. Και σύμφωνο με τον κύριο Τεγιόγκ ότι οι Ιταλοί έχουν μια καταπληκτική νομοθεσία και ίσως την καλύτερη νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα αυτό. Βέβαια, ναι, και οι Ολλανδοί έχουν καλή νομοθεσία και στην Ιταλία έχουν και πολλές επιτροπές ε, και πολύ καλή άρτια νομοθεσία, αλλά παρόλα αυτά το φαινόμενο της μαφίας δεν έχει εξαλειφθεί παρά τις προσπάθειές τους ε, ε, τα τελευταία δέκα χρόνια εξακολουθεί να ελιμένεται η, Ιταλία, η μαφία την Ιταλία. Τι πήγε στραβά λοιπόν, πού χωλένει η κατάσταση. Κανονικά η Ιταλία θα πρέπει να ήταν απαλλαγμένη μετά από τόσες μακροχρόνιες προσπάθειες από τη μαφία. Είπε ο κύριο ε, ε, είναι τον Νταν, μήπως κάναμε διαφήμιση στου Ιταλού. Ε, ε, ίσως ήταν ένα, μια παράπλευρη συνέπεια, αλλά Τώρα που έκλεισε το θέμα, ίσως σκόπιμο θα ήταν να πάμε και σε άλλες χώρες. Είδατε τις μελέτες που έγιναν στη Γερμανία, στην Ιταλία και οι χώρες αυτές κατηγορήθηκαν ότι δεν κάνουν αρκετές προσπάθειες για την πάταξη της ε, διαφθοράς. Ε, λιγότερο μιλάμε για τις χώρες αυτές ε, που δεν έχουν πολύ αυστηρές νομοθεσίες κατά της διαφθοράς. Και έτσι τη γλιτώνουν αυτές οι χώρες ελάχιστα αναφέρονται. Βέβαια μπορεί να μην υπάρχει μαφία σε αυτές τις χώρες με τα χαρακτηριστικά της Ιταλίας, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει διαφθορά. Να μην επικεντρωθούμε μόνο στην Ιταλία. Μπορεί στις άλλες χώρες να μην είναι τόσο θεαματική η δράση των παράνομων οργανώσεων όπως της μαφίας στην Ιταλία, αλλά και εκεί έχουμε πολλά φαινόμενα και καλό θα ήταν και οι άλλες χώρες να μας απασχολήσουν που μέχρι, στιγμές, μέχρι στιγμής έχουν μείνει στην ανωνυμία. Γιατί στην Ιταλία πολύ θόρυβος γίνεται και πάταγος, αλλά αποτελέσματα δεν βλέπουμε και πολλά τελικά. Ο κύριος Σόρενγκατ, ε, μετά θα ακούσουμε την παρουσίαση του κυρίου De Jong για τη διαφθορά στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και να δώσω το λόγο στην κυρία Βάιλερ. Δύο σύντομες απαντήσεις. Ε, ναι, έχετε δίκιο κύριε συνάδελφε. Το ίδιο θα πρέπει να συμβεί και στη Γερμανία και στην Γαλλία. Γιατί στη Γερμανία υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Και νομίζω ότι αυτές είναι οι δύο πιο μεγάλες ε, χώρες που, κάνουν, ε, που σαν να ήταν τα πράγματα, σαν να ήταν όλα εντάξει. Στον, ε, προς τον Δανό συνάδελφο. Κατά την άποψή μου υπάρχουν δύο λόγοι γι' αυτό. Το πρώτο είναι η αλλαγή της μαφίας. Η μαφία είναι ισχυρότερη από ποτέ. Έστω και αν ε, υπάρχει κάποια κοινωνική επαξίωση, τουλάχιστον στην Νότια Ιταλία, έναντι της μαφίας. Δηλαδή δεν τρέμουν όλοι ε, μόλις εμφανιστεί η μαφία. Αλλά έχει αλλάξει πρόσωπο η μαφία. Ε, και μέσω διαφόρων ε, ε, ε, από, από, το, από τη λέξη η οποία δούλευε κάνοντας ε, δολοφονίες τελικά μεταμορφώθηκε σε μια ευυπόλυπτη ομάδα η οποία συμμετέχει σε ξέπλυμα χρημάτων και σε, άλλου είδους, σε κάποιες εγκληματικές ενέργειες αλλά χωρίς να κάνει άμεσα δολοφονίες ή φανώσω ε, κατά την άποψή μου στην Ιταλία τα πράγματα είναι δύσκολα γιατί υπάρχει διαπλοκή με την πολιτική. Νομίζω αυτή είναι η απάντηση. Ε, Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι αυτή η σύντομη συζήτηση που είχαμε μας άνοιξε την όρεξη για να διαβάσουμε τις 30 σελίδες, την διεξοδική παρουσίαση δηλαδή των ε, τεκτενωμένο στην αντιπροσωπεία και την αποστολή της αντιπροσωπείας μας στην Ιταλία, στις τρεις αυτές πόλεις. Μπορούμε λοιπόν να διαβάσουμε αυτή την λεπτομεριακή έκθεση που περιλαμβάνει και τις προτάσεις και διάφορα στοιχεία των διάφορων συνομιλητών μας στην Ιταλία και στοιχεία για τις τοσελίδες τους. Είναι πολύ πλούσια και εξονυχιστική αυτή η έκθεση από την αποστολή στην Ιταλία και σας έχει μοιραστεί. Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, που είναι το κυρίως θέμα της σημερινής μας συζήτησης και που προβλέπει την παρουσίαση και συζήτηση για τέσσερα για τέσσερις θεματικές ενότητες και αντίστοιχα έγγραφα με θέμα τη διαφθορά. Σε αυτά τα τέσσερα thematic papers, όπως τα λέμε στα αγγλικά, περιλαμβάνονται διάφορες προτάσεις και πολλά στοιχεία τους αναφέρονται και στην ε, έκθεση, στο έγγραφο εργασίας του εισηγητού μας η οποία έχει αποστολή για, τη μετα... για μετάφραση. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η μετάφραση. Ε, η συζήτηση του εγγράφου εργασία του εισηγητού θα γίνει τον Ιανουάριο, μέχρι όταν ολοκληρωθεί και η μετάφραση του εγγράφου. Αλλά έχετε λάβει στα αγγλικά το σημείο με της γραμματείας για τα τέσσερα αυτά θεματικά έγγραφα. Το έγγραφο εργασίας, επαναλαμβάνω, θα το εξετάσουμε τον Ιανουάριο. Τώρα θα ακούσουμε τους συντάκτες των τεσσάρων ε, θεματικών ε, ενωτήτων για τη διαφθορά. Το πρώτο θέμα θα παρουσιαστεί από την κυρία Μαρία Καμπριέλ για τη διαφθορά στις δημόσιες προμήθειες. Μετά θα έχουμε τα ευρωπαϊκά ταμεία και τη χρήση τους από το, κατάχρηση τους από το οργανωμένο έγκλημα. Παρουσίαση της κυρίας Βάιλερ. Το τέταρτο έγγραφο αφορά ε, τομείς ε, συστημικής διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση των κρατών μελών και μέτρα για να καταπολεμηθούν τα αρνητικά τη αποτελέσματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριο Θαδός Κυλακάκη από την Άλντε είναι ο συντάκτη αυτού του εγγράφου και τέταρτο έγγραφο ε, αφορά τη διαφθορά στι ιδιωτικέ επιχειρήσει που διαταράσσουν το θεμητό ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Ο κύριος Δεγιόνκα από την ΚΟΕ είναι ο συντάκτης αυτού του τέταρτου εγγράφου. Προτείνω για τη συζήτηση να δώσουμε σε κάθε συντάκτη 15 λεπτά για την παρουσίαση του εγγράφου του και θα σας χειροκροτήσουμε ακόμη περισσότερο αν περιοριστείτε σε ακόμη λιγότερο χρόνο, δεν εξαντλήσετε δηλαδή το 15 λεπτό, ώστε να έχουμε μία ώρα για να συζητήσουμε μετά τα τέσσερα θεματικά έγγραφα. Θα, στη συζήτηση θα δοθεί προτεραιότητα ε, φυσικά στον εισηγητή, στους ε, εκπροσώπους και συντονιστές των πολιτικών ομάδων και μετά θα ακούσουμε και τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μας παρουσιάσει το δικό της έργο σε θέματα πάταξης της διαφθοράς. Οπότε μετά από το γύρο της συζήτησης ε, για τα έγγραφα αυτά θα ακούσουμε και τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και φυσικά θα δευτερολογήσουν οι συντάκτες των εγγράφων. Θα ξεκινήσουμε από το πρώτο έγγραφο που αφορά τη διαφθορά στις δημόσιες προμήθειες. Η Μαρία Γκαμπριέλ είναι η συντάκτη του πρώτου αυτού εγγράφου. Παρακαλώ, σας ακούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να παρουσιάσω αυτό το θεματικό έγγραφο ε, με τιμά ιδιαίτερα το καθήκον αυτό. ασχολείται με ένα πολύ σημαντικό θέμα, τη διαφθορά και μάλιστα στις δημόσιες προμήθειες, γιατί ξέρουμε ότι οι κρατικές προμήθειες ε, συνάπτονται μεταξύ των δημοσίων αρχών και ιδιωτών ή δημόσιων φορέων. Είναι πολύ ε, επιρρεπής τομέας αυτός ε, στη διαφθορά. Οπότε είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να μεριμνήσει ώστε οι δημόσιες προμήθειες να είναι διαφανείς και ανοιχτές προς το ευρύ κοινό. Στο εγγραφό μου ε, καταρχήν ασχολήθηκα με το θέμα των ορισμών. Στο πρώτο τμήμα λοιπόν του εγγράφου ε, μιλάω για τη δυσκολία ε, συμφωνίας σε ένα κοινόρισμό. Ε, στη συνέχεια έκανα μια σύντομη επισκόπηση των διαφόρων νομοθεσιών, διεθνών και ευρωπαϊκών και με βάση την ανάλυση και της ε, κοινωτικής νομοθεσίας θα υποβάλουμε και κάποια συμπεράσματα στο τρίτο σκέλος του εγγράφου. Χρειαζόμαστε ένα στέρεο νομικό πλαίσιο και μια σωστή εφαρμογή της ε, νομοθεσίας. Θα πρέπει όμως εξ αρχής να πούμε ότι είναι δύσκολο να δώσουμε στατιστικά στοιχεία για όλες τις ζημίες οικονομικές και δημοσιονομικές που προκαλούνται από την ύπαρξη της διαφθοράς στις ε, δημόσιες προμήθειες. Δεν ε, εντοπίζονται εύκολα όλες αυτές οι ζημίες και δεν μπορούν να αποτιμηθούν κιόλα τα στατιστικά, θα τα στατιστικά στοιχεία θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να καταλήξουμε σε ένα σύστημα κοινών δικτών για να επικεντρωθούμε περισσότερο στην πρόληψη. Χαιρετίζω πάντως ιδιαίτερα την ε, πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να θεωρηθεί το νομικό πλαίσιο για τις δημόσιες προμήθειες. Έτσι θα ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στα κοινοτικά θεσμικά όργανα και θα ενταθούν οι προσπάθειες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών για να παταχθεί η διαφθορά ή να καταπολεμηθεί με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Η πρώτη δυσκολία έγκυται στην έλλειψη του κοινού ορισμού. Αναφέρεται ο ορισμός των Ηνωμένων Εθνών για τη διαφθορά, που τη χαρακτηρίζει ως φαινόμενο που απειλεί τη σταθερότητα και την ασφάλεια των κοινωνιών, υπονομεύει τα θεσμικά όργανα και τις δημοκρατικές ηθικές αξίες και τη δικαιοσύνη, και που διακυβεύει την αηφόρο ανάπτυξη και το κράτος δικαίου. Έχουμε όμως και δύο άλλους ορισμούς, που είναι ο ορισμός του ΩΣΑ, αλλά έχουμε και τον ορισμό της Transparency International, της διεθνούς διαφάνειας. Η διεθνή διαφάνεια τονίζει ότι η διαφθορά στις δημόσιες αγορές καλύπτει ε, τη, διαφθορά, τη σύγκρουση ε, συμφερόντων και την καταβολή προμηθειών διαφθορά λοιπόν φτάνει, ε, αγγίζει και τα πέντε επίπεδα, την αξιολόγηση, την προετοιμασία, η επιλογή των προμηθευτών, ε, των, ε, προμηθευτών των προϊόντων, ε, το λογιστικό θέμα και το θέμα της πρόληψης. Θα πρέπει λοιπόν να εντοπίσουμε τα διάφορα στάδια στα οποία μπορεί να εμφανιστεί η διαφθορά και στα πλαίσια αυτά ασχοληθήκαμε και με την παγκόσμια και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπουν τα θέματα αυτά. Σε διεθνές επίπεδο ε, διαπιστώσαμε ότι τρία είναι τα σημαντικά έγγραφα που ε, θεσπίζουν αυτό το νομικό πλαίσιο. Έχουμε καταρχήν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς που είναι το πιο σημαντικό νομικό έγγραφο. 140 χώρες έχουν υπογράψει και κυρώσει αυτή την ε, σύμβαση του ΟΗΕ και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εξαίρεση την Γερμανία και την Τσεχία που ποτέ δεν ε, κύρωσαν την έκθεση. Επίσης έχουμε την σύμβαση του ΟΣΑ για την καταπολέμηση της, αυθοράς, ε, της διαφθοράς στις ε, διεθνείς εμπορικές συναλλαγές. Η σύμβαση αυτή μας προσφέρει κάποια νομικά μέτρα και τρόπους για να καταπολεμηθεί η διαφθορά στις δημόσιες προμήθειες ενώ και τα κράτη του G20 το 2010 υιοθέτησαν ένα σχέδιο δράση για την καταπολέμηση διαφθορά. Τρίτο στοιχείο είναι η Συμφωνία για τι Δημόσιε Προμήθειε, μια διεθνή συνθήκη υπό την αιγίδα τη Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου, ένα άλλο πολύ σημαντικό δηλαδή νομικό έγγραφο συμφωνήθηκε από 42 χώρες, μεταξύ των οποίων είναι και 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφού λοιπόν κάναμε μια επισκόπηση της διεθνούς νομοθεσίας, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει πρόβλημα μεταξύ της ύπαρξης των νομικών κειμένων αφενός και της εφαρμογής του αφετέρου. Ε, στη συνέχεια ασχοληθήκαμε με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα θέματα αυτά. Διαπιστώσαμε ότι αφενός οι συνθήκες ε, προβλέπουν μια γενική νομική βάση για το θέμα αυτό, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και δύο οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ε, τις δημόσιες προμήθειες. Η πρώτη είναι η οδηγία που αφορά τις δημόσιες προμήθειες για έργα, ε, προμήθειες και υπηρεσίες και η δεύτερη οδηγία είναι την ε, ανάθεση συμβάσεων για το είδωρ, ενέργεια, μεταφορές και ταχυδρομικές υπηρεσίες. Οι οδηγίες αυτές το έχουν την εξασφάλιση του ανοίγματο ε, των προμηθειών στην, ε, στην, στον ανταγωνισμό, προκειμένου να εξασφαλιστεί ελεύθερη και χωρί διακρίσει πρόσβαση των επιχειρήσεων στι δημόσιε προμήθειες. Παρά όμω στο νομικό αυτό πλαίσιο, διαπιστώνουμε ότι η διαφθορά στι δημόσιε προμήθειες δεν αποτελεί δυστυχώ την εξαίρεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι, προκειμένου να αναθεωρήσουμε το νομικό σύστημα αλλά και να καλύψουμε κάποια νομοθετικά κενά. Χαιρετίζουμε τις τρεις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υπευλήθησαν το 2011. Έτσι, τα θεματικά αυτά έγραφα αφιερώνουμε ένα σημαντικό τμήμα στην ανάλυση των προτάσεων της Επιτροπής του 2011. Καταρχήν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την, έκθεση, την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για τις δημόσιες προμήθειες. Και μάλιστα έχουμε και την πρόταση αυτή που αφορά τις ε, δημόσιες προμήθειες ε, για το είδωρ ενέργεια, ε, μεταφορές και ταχυδρομικές υπηρεσίες. Στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε οδηγία για τις συμβάσεις παραχώρησης, που μέχρι στιγμής μόνο μερικά διαθετούνταν και φέτος δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα έγγραφο εργασίας το οποίο κάνει μια αξιολόγηση της υφιστάμενης νομοθεσίας. Για παράδειγμα, στο έγγραφο αυτό αναφέρονται ότι μόνο εννέα χώρε έχουν εσωματώσει την ιστορική του νομοθεσία την οδηγία για τι δημόσιε προμήθειε και μάλιστα εμπρόθεσμα, εγκαίρω. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε και το ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι ένα ρόλο εποπτεία, εξακρίβωση τη σωστή εφαρμογή τη κοινοτική νομοθεσία και τη σωστή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Αλλά επειδή δεν υπάρχει κοινό σύστημα, δεν μπορεί να κάνει μια πλήρη και εμπεριστατωμένη επισκόπηση της κατάστασης στα κράτη-μέλη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι οι δημόσιε προμήθειε είναι ιδιαίτερα ευάλωτε ε, και, ε, και στην απάτη αλλά και στην κατασπατάληση των δημοσίων πόρων και για να καταπολεμηθεί η διαφθορά στις δημόσιες προμήθειες ε, θα δύο σημαντικές συστάσεις. Οι συστάσεις αυτές όμως ε, δικαιολογούνται από πολύ συγκεκριμένες αρχές. Χρειαζόμαστε περισσότερη διαφάνεια, ενισχυμένο νομικό πλαίσιο, ανοιχτού διαγωνισμού, ένα σύστημα ηλεκτρονικό για τη σύναψη, επίση ε, προστασία των καταγγελόντων και ένα κοινό σύστημα εποπτείας και επιτήρησης. Χάρη στι ε, αρχές αυτές θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε δύο σημαντικέ προτεραιότητε που θα πρέπει να εφαρμοστούν μέσω και μακροπρόθεσμα. Καταρχήν ε, να καταρτήσουμε ε, συγκεκριμένους ε, κοινούς δείκτες και ένα σύστημα συναγερμού που είναι απαραίτητο για το, για το σύστημα εποπτείας μας και να καταλήξουμε σε συγκεκριμένο προσδιορισμό των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων σε ό,τι αφορά την επιτήρηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτές οι δύο συστάσεις είναι μέτρα που καλό θα ήταν να θεσπιστούν και να εφαρμοστούν και εμπράκτορος ώστε να στείλουμε ένα χειρό μήνυμα και προς τις δημόσιες διοικήσεις αλλά και προς τους Ευρωπαίους πολίτες και θα ήθελα να πω ότι πιστεύω ακράδαντα πως ο ένας από τους καλύτερους τρόπους για να ελαχιστοποιήσουμε τη διαφθορά είναι να ε, μελετήσουμε διεξοδικά αυτό το θέμα, να καταρτήσουμε κάποιες προτεραιότητες, να δούμε ποιες δράσεις θα πρέπει να λάβουμε και φυσικά να καταλήξουμε σε κοινή προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να καταπολεμηθεί αυτή η μάστιγα. Όλα αυτά αναφέρουμε στο θεματικό έγγραφο. Σας παρουσίασα την δομή. Έχουμε πρόβλημα λόγω έλλειψης κοινού ορισμού. Κάναμε μια επισκόπηση της υφιστάμενης νομοθεσίας. Προσκρούσαμε στο πρόβλημα που υπάρχει με τη διαφάνεια, την εφαρμογή Γι' αυτό και ζητούμε ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο και κάποιες τεχνικές διατάξεις ώστε να ανοίξουν πραγματικά οι αγορές και νομίζω ότι οι δύο συγκεκριμένες μας συστάσεις αφορούν τα απαραίτητα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν βράχη και μέσο πρόθεσμα ώστε να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε και τον απότερο μας στόχο που είναι η πλήρης εξάλληψη της διαφθοράς στις δημόσιες προμήθειες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Καμπριέλ πολύ εμπεριστατωμένη και διεξοδική παρουσίασή σας και ήδη διαμορφώσαμε μια ιδέα για τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που μας περιμένουν. Μάλιστα προλάνεται το έδαφος και για τη δεύτερη παρουσίαση που είναι το θεματικό έγγραφο της κυρίας Βέιλερ για τα ευρωπαϊκά ταμεία και την κατάχρηση που γίνεται από το, διεθνές, από το οργανωμένο έγκλημα. Äh, Ωραία λοιπόν. το θέμα αυτό, το πώς η οργανωμένη εγκληματικότητα χρησιμοποιεί, εκμεταλλεύεται τα ευρωπαϊκά ταμεία. Εδώ έχουμε ακόμα μεγαλύτερες ε, δυσκολίες να εξεύρουμε δεδομένα γιατί πραγματικά αυτό ε, συμβαδίζει με τη φύση του πράγματος, δηλαδή θα πρέπει όλα να μείνουν ε, μυστικά. Και όσον αφορά το δίκαιο ανάθεση δημόσιων έργων, εδώ έχουμε την ε, τύχη ε, οι υποψήφοι οι οποίοι απορρίπτονται προσφεύγουν ορισμένες φορές και λένε ότι δεν έχουν, γίνει, δεν έχουν τύχει σωστή μεταχείριση. και άρα υπάρχει μια υπηρεσία που οποία ε, ασχολείται με αυτά τα στοιχεία. Ε, τώρα, όσο, επίσης ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι όσον αφορά τα διορθωτικά τομεία, όταν πρόκειται για οργανωμένη εγκληματικότητα και όχι για απλά φαινόμενα απάτηση ε, ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μεγάλη κατάτμιση ε, και ε, σπορά των αρμοδιοτήτων, κατάτμιση των αρμοδιοτήτων και διάφοροι τομείς που ασχολούνται με την καταπολέμηση του εγκλήματος. Στο δικό μου κείμενο προσπάθησα στην αρχή να διατυπώσω έναν ορισμό. Δεν υπάρχει ένας επίσημος έγκυρος ορισμός, αλλά εμεί επιχειρήσαμε να κάνουμε, να σε έναν ορισμό. Δηλαδή είπαμε ότι η οργανωμένη, το οργανωμένο έγκλημα είναι μια ένωση, μια διαφωμένη ένωση η οποία ε, αν βρει μια μορφή συνεργασία για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, πρέπει να είναι πάνω από δύο άτομα τα οποία συμμετέχουν εδώ και βεβαίω θα πρέπει να διαπράττουν κάποιε αξιόπινε πράξει, να πληρούν κάποια σχετικά κριτήρια. Για παράδειγμα, ε, που να αντιστοιχούν σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση, ανάλογα με το ποιο είναι το προβλόμενο σύστημα του κάθε κράτους. και υπάρχει ο στόχος να ε, αποκομίσουν ένα οικονομικό ή άλλο όφελος από αυτό το εγχείρημα. Ε, τα γνωρίζετε όλα αυτά, όλα αυτά τα έχω συμπεριλάβει σε έναν κατάλογο ε, ποια είναι τα οικονομικά συμφέροντα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οικονομικά της έσοδα Ε, τα διάφορα ποστά 1,1% ή 1,9% ανάλογα με το πόσο καταβάλουν τα κράτη-μέλη. Ε, επίσης τα έσοδα από διάφορα μεγάλα καρτέλ, συγχωνεύσεις. Ε, οι σημαντικότερες μορφές απάτης είναι η απάτη σε σχέση με το ΦΠΑ και με το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Αυτά είναι... Από εδώ προέρχονται τα μεγαλύτερα έσοδα. Και επίσης ε, προσπάθησα στο κείμενό μου να εξηγήσω ή να διευκρινίσω ότι είναι δύσκολο να διακρίνουμε, να κάνουμε μια διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων και επίσης είναι δύσκολη δίωξη γιατί δεν έχουμε ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό σύστημα εδώ και αυτό θέλουμε να το επεξεργαστούμε. Έχουμε μεν μια οδηγία για το ξέπλυμα των χρημάτων και έχουμε μια οδηγία εδώ ε, τάπητος ε, σε σχέση με τι θα πρέπει να γίνει με τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία αλλά τελικά αυτά εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο από τις, εθνικές, από τις αρμόδιες εθνικές αρχές και όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η... Ο έλεγχος ε, η εξέταση μάλλον του τι είναι οργανωμένη εγκληματικότητα και πού διαπιστώνονται τέτοια φαινόμενα, ή τέτοια περιστατικά. Είναι δύσκολο να διεξαχθεί αυτός ο έλεγχος γιατί ε, οι χώρες μέλη που κάνουν κάτι τέτοιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση από την άλλη ε, έχουν εντελώς διαφορετικού διαφορετικούς πόρους. Και τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν τους οικονομικούς πόρους για να προβούν σε κάτι τέτοιο. Για παράδειγμα, στην Ιταλία, ε, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούσε να κάνει αυτό το οποίο κάνει η Ιταλία. Δεν έχει καν το αντίστοιχο προσωπικό, το αναγκαίο προσωπικό. Ε, εδώ υπάρχουν ορισμένες οργανώσεις ε, που υποβοηθούν και σε αυτές συγκαταλέγεται και η Όλαφ. Η Europol και η Eurojust είναι οι άλλες ε, υπηρεσίες. Αυτές νομίζω είναι οι τρεις βασικές υπηρεσίες που αναλαμβάνουν εδώ ένα ενεργό ρόλο και εμείς ε, είμαστε ιδιαίτερως εξαρτημένοι από την ανάλυση της Όλαφ. Η Όλαφ έχει καταγράψει κάποιες τέτοιες περιπτώσεις και πρόκειται να τις δημοσιεύσει και διαπιστώνει ότι υπάρχει μια αύξηση αυτών των περιπτώσεων και στο επίπεδο των χωρών μελών, για παράδειγμα στη Γερμανία έχουν αυξηθεί αυτά τα φαινόμενα. Εγώ στην παρουσίασή μου δεν αναφέρω τους πολιτικούς λόγους, γιατί ασφαλώς ε, προσεγγίζω διαφορετικά από την κάθε πολιτική ομάδα, αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτή η αύξηση της ε, απάτης Συναντάται βεβαίω στενά με την ε, χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία έχει ε, εμφανίσει επιπτώσει σε όλες τις ε, χώρες μέλη και η οποία βεβαίως αυτές τις ενθαρρύνει υποστηρίζει αυτές τις ομάδες που ασκούν, που κάνουν τις απάτες, τους παροτρύνει, τους μάλλον δίνει ένα κινήτρο να κάνουν αυτές τις εγκληματικές ενέργειες. Στην Ιταλία ε, είναι εξόφθαλμο το γεγονό ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια γίνονται αντικείμενο μια ιδιαίτερη εκμετάλλευση, ιδιαίτερα μεγάλη εκμετάλλευση. Και εκτιμώ ότι αυτό θα συμβαίνει και σε κάποιες ε, από τις πιο καινούριε χώρε μέλη από την ε, Ανατολική Ευρώπη. Αλλά αυτό δεν είναι αναγκαστικό. Για παράδειγμα, η δική μου χώρα, σαν αφορά για παράδειγμα στη Βαυαρία, Υπάρχουν τέτοια περιστατικά όπου καμιά φορά κανείς κινείται σχεδόν στο όριο του να ορίσει κατά πόσο πρόκειται για μεμονωμένα άτομα ή πράγματι για μορφές οργανωμένης εγκληματικότητας από σπήρες. Είναι σχετικά σπάνιο να κάνει τις απάτες μια πραγματικά οργανωμένη σπήρα. Και αυτό ιδιαίτερο αφορά τα μέτρα των, τα, τα, τα, μεγάλα έργα, τις υποδομές, τη δημιουργία ε, δρόμων, ε, εγκαταστάσεων ε, καθαρισμού αυτοκινητοδρόμων κλπ. Εδώ γίνονται οι περισσότερες απάτες και ίσως εδώ η Κομισιόν θα πρέπει να θεσπίσει άλλες μεθόδους ή όργανα για να μπορέσει να διαπιστώσει κατά πόσο τα, να έχουμε κάποια ευρωπαϊκά κονδύλια από τα διευθυντικά ταμεία. Ε, ε, Βεβαίω, είναι λίγα αυτά τα πολύ μεγάλα προγράμματα ε, και θα πρέπει να είναι προσεκτική η Κομισιόν ευθύς εξ αρχής νομίζω από την αρχή της ανάθεσης του έργου μέχρι την, όλη την πορεία της υλοποίησής του. Και εδώ στον κατάλογο μου περιλαμβάνω ένα project το οποίο έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο πλαίσιο αυτό το project Καπάτσι στην Ιταλία. Όποιος ε, συμμετείχε εδώ στην Ενδράση τη Επιτροπή έχει μια αντίληψη περί τίνο πρόκειται εδώ. Ε, αυτό το πρόγραμμα υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει μια παρακολούθηση, ένα monitoring για τα μεγάλα δημόσια έργα και όπου η ροή, ε, οι χρηματοοικονομικές ροές ε, μεταξύ των διαφόρων ε, τραπεζών εξετάζονται επακριβώς. Γιατί πολύ συχνά διαπιστώνονται εδώ κάποια περιστατικά ξεπλήματος χρημάτων. Και θα δούμε τι θα γίνει όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα αυτό. Θα δούμε δεχομένω ποια είναι τα αποτελέσματα και θα υπάρξει μια σχετική ακρόαση. Λοιπόν, θα έρθω τώρα στα συμπεράσματα και ε, στα αιτήματα τα οποία κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να θέσει η δική μας Επιτροπή με το μέσω του βασικού εισηγητού αλλά και μέσω των άλλων ενδιαφερόμενων αρμοδίων επιτροπών. Καταρχήν το επίπεδο της πρόληψης, γιατί έχουμε την εντύπωση ότι στο επίπεδο αυτό δεν γίνονται αρκετά πράγματα. Βεβαίω ε, αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει. Χρειαζόμαστε ιδιαίτερως ε, πεπειραμένους ειδικού ή εξωματούχους υπαλλήλους που έχουν μια σχετική εμπειρία ενδεχομένω το πού θα μπορούσαν να πάνε στραβά τα πράγματα. Η λοιπόν, σημαντική εδώ. Και επίση Και επίση θα ήθελα να φέρω αυτό που πολλοί συνάδελφοι ειναι ιδιαιτερω σημαντικη εδω και επίση θα ηθελα να φέρω αυτο που πολλοι συναδελφοι εχουν συμπελαβει και στου παρουσιάσει, μια, δηλαδή μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μια Ευρωπαϊκή Διοκτική Αρχή, γιατί ε, πραγματικά η διαπλοκή στις διάφορες ε, ε, όχι, η σχέση μεταξύ μάλλον των διαφόρων χωρών, ποια χώρα κάνει τι, η Αυστρία, η Ιταλία, η Γερμανία κλπ. Όλα αυτά δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, αλλά μπορούμε τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο να θεσπίσουμε ένα δεσμευτικό πλαίσιο με κάποιες δεσμευτικές ρυθμίσεις. Και επίσης οι χώρες μέλη θα πρέπει να κάνουν περισσότερα πράγματα όσον αφορά τις απάτες με το ΦΠΑ και το λαφρεμπόριο τσιγάρων και το λέω ξεκάθαρα γιατί ε, βλέποντας ε, όλες τις ιστορίες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το κοινοβούλιο ο, τι αγώνες πρέπει να κάνουμε γύρω από τον προπολογισμό για να μπορέσουμε να παγιώσουμε συστηματικά τέτοιε προσπάθειε. Γιατί νομίζω ότι όλες οι πολιτικές ομάδες παλεύουν με το Συμβούλιο για κάτι τέτοιο. για τον προπολογισμό, αλλά όταν γίνεται, αν γινόταν μια εξίσου συστηματική προσπάθεια σχέση με την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, νομίζω ότι θα μπορούσαμε εύκολα να είχαμε σημειώσει πρόοδους. Ένα άλλο σημείο είναι οι συμφωνίες με τις τρίτες χώρες, με το Λίχτενστάιν, με την Ελβετία κάναμε κάποια πράγματα, με το Λίχτενστάιν δεν έχει ακόμα ψηφιστεί νομίζω ότι όλα αυτά περιλαμβάνουν πράγματα που εμεί θεωρούμε σημαντικά. Αυτά είναι τα σημεία τα οποία ήθελα να επισημάνω και θα ήθελα κλείνοντα να σα ευχαριστήσω γιατί πραγματικά πολύ ουσιαστική βοήθεια τη Γραμματεία. Σα ευχαριστούμε κυρία Βάιλερ για την παρουσίαση του εγγράφου διαφθορά στη χρήση των ταμείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το οργανωμένο έγκλημα θα πρέπει να γίνει κάποιος έλεγχος ε, των δαπανών ε, σε θέματα υποδομής ε, και να χρησιμοποιήσουμε τους μηχανισμούς που έχουμε όπως η ΟΛΑΦ που έχει σημαντικές αρμοδιότητες, ακόμη και οι υποκλοπές, παρακολουθήσει τηλεφωνικών συνομιλιών κλπ. Και φυσικά θα πρέπει να ασκήσουμε και εμείς τον κοινοβουλευτικό μας έλεγχο. Πέραν των θεμάτων της ποινική δικαιοσύνη, που θα συζητηθούν σε μια ειδική δημόσια κρόαση που θα γίνει την εβδομάδα αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άλλωστε, σε αυτά τα θέματα αναφέρεται και η έκθεση De Jong, έκθεση πρωτοβουλίας που θετήθηκε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πριν όμως δώσουμε το λόγο στον κύριο De Young, θα ακούσουμε το άλλο πολύ σημαντικό θεματικό έγγραφο για ένα θέμα που απαιτεί τη συνεργασία μεταξύ των διοικήσεων των κρατών μελών για να καταπολεμηθεί η διαφθορά το θεματικό έγγραφο του κυρίου Σκυλακάκη και αυτό το θέμα αφορά το θέμα της συστημικής διαφοράς της δημόσιας διοίκησης των κρατών μελών και ποια μέτρα είναι απαραίτητα να εφαρμοστούν προκειμένου να παταχθεί το αρνητικό αποτέλεσμα αυτής της συστημικής διαφθοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δώσω λοιπόν αμέσως το λόγο στον συνάδελφό μας, τον κύριο Σκυλακάκη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω αναφέροντας ότι η, διαφορά, ε, η δυσκολία με τη διαφθορά είναι ότι είναι δύσκολα μετρήσιμη. Δηλαδή οι άνθρωποι αισθάνονται, το διαισθάνονται ότι η διαφθορά είναι ευραίως διαδομένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πρέπει να πω ότι δεν έχουμε δει συγκεκριμένα στοιχεία για το πώς ακριβώς προσμετράται αυτή η διαφθορά. Η Transparency International μας έχει δώσει κάποια στοιχεία, τα οποία όμως κατά την άποψή μου δεν έχουμε εξετάσει ενδελεχώς. Γι' αυτό λοιπόν εγώ προέβηνε σε μία ανάλυση αυτών των δεδομένων, όπου οι άνθρωποι οι ίδιοι λένε ότι δηλώνουν σε σφιγμομετρήσεις ότι δωροδόκησαν κάποιον σε ένα συγκεκριμένο τομέα, δημόσιο τομέα. Εδώ και χρόνια γίνονται έρευνες από αυτού για πολλές χώρες ε, και στην Ευρώπη και εκτός αυτής. Εάν λοιπόν σε μία και μόνο χρονιά κάνουμε το άθροισμα των οικοκυριών όπου κάποιος έχει δωροδοκίσει έναν δημόσιο υπάλληλο σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα, τότε καταλήγουμε σε περίπου 20 εκατομμύρια δωροδοκίες ανά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επαναλαμβάνω τα στοιχεία, γιατί δεν το συλλαμβάνει κανείς εύκολα τον αριθμό αυτό, 20 εκατομμύρια δωροδοκίες απλών πολιτών ε, γιατί προφανώ σε, σε μια έρευνα δεν μπαίνει κανεί σε έναν επώνυμο πολιτικό να τον ρωτήσει δωροδοκηθήκατε και να πει αυτό μάλιστα ναι, σωστά, δωροδοκήθηκα. Απλών λοιπόν πολιτικών, ε, πολιτών, με συγχωρείτε. Αυτό λοιπόν πρώτα απ' όλα πρέπει κανείς να συλλάβει. Και αυτά είναι τα ελάχιστα στοιχεία. Αυτό μας το λένε οι ίδιοι οι πολίτες. Δεν είναι τι πιστεύουμε ή εικάζουμε ότι έχει γίνει. Οι πολίτες καταθέτουν ότι αυτό έγινε. Και δεν το λένε έτσι γενικά και όριστα, το αναφέρουν πολύ συγκεκριμένα. Γνωρίζουμε λοιπόν, ε, με βάση τα νοικοκυριά που απάντησαν, ότι περίπου 600.000 νοικοκυριά στην Ευρώπη δήλωσαν ότι έχουν δορδοκίσει τα τελωνία, τις τελωνιακές αρχές. Ε, αναφέρομαι στις τελωνιακές αρχές γιατί αυτές ε, παίζουν σημαντικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση από πλευράς οικονομικής ίσπραξης χρημάτων. Ε, εμείς ε, δεν ξέρουμε βέβαια συγκεκριμένους αριθμούς, ε, δεν θέλουμε όμως δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις να μάθουμε τους πραγματικούς αριθμούς, γιατί αν το κάνουμε αυτό τότε θα πρέπει και κάτι να κάνουμε. Αυτό, αυτή τη δυσκολία ενέχουν οι αριθμοί. Ας δούμε τώρα ποιες είναι οι επιπτώσεις. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οφείλω να σας πω ότι ε, ποικίλουν τα στοιχεία πάρα πολύ ανατομέα και αναχώρα. Υπάρχουν χώρες, δεν θέλω τώρα να τις ονοματίσω, όπου σε πάρα πολλούς τομείς έχουμε μηδενική διαφθορά και άλλες πάλι χώρες όπου το 30% των πολιτών κάθε χρόνο προβαίνουν σε πράξεις δωροδοκίας σε συγκεκριμένους τομείς. Παραδείγματο χάρη, στον τομέα των δημόσιων νοσοκομείων διαπιστώνουμε εκτεταμένη διαφθορά σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Τώρα, αν το ονοματίζουμε ως διαφθορά ή όχι, σημασία έχει ότι καταβάλλονται ε, φακελάκια στους ε, γιατρούς ε, για υπηρεσίες που θα έπρεπε έτσι και αλλιώς να έχουν προσφέρει στο δημόσιο τομέα. Πάντως αυτό το φαινόμενο επεκτείνεται και σε άλλους τομείς. Εφόσον λοιπόν είναι τόσο ευρέως διαδεδομένη η διαφθορά, πώς πρέπει να την αντιμετωπίσουμε και πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Ας δούμε πώς επηρεάζει τα οικονομικά συμφέροντα καταρχήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τομείς από τους οποίους συλλέξαμε πληροφορίες, αυτοί δεν σχετίζονται άμεσα με οικονομικά συμφέροντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξαιρουμένων των τελωνίων. Αν όμως γνωρίζει κανείς ότι η διαφθορά είναι διαδεδομένη στη δημόσια διοίκηση και σε τελική ανάλυση ε, είναι οι ίδιοι υπάλληλοι που ε, δωροδοκήθηκαν σε εθνικό επίπεδο και αυτοί χειρίζονται τα κοινοτικά κονδύλια, καταλαβαίνετε ε, την έκταση του φαινομένου. Παραδείγματο χάρη, οι γεωργοί αυτοί δεν ερωτώνται ποτέ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει κάνει έρευνες σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, κάτω από το πρίσμα εκείνων που εμπλέκονται ουσιαστικά σε τέτοιου είδου υποθέσεις. Άρα δηλαδή δεν γνωρίζουμε, αλλά μπορούμε να εικάσουμε ότι η διαφθορά είναι πολύ περισσότερο διαδεδομένη από αυτό που πραγματικά βλέπουμε. Ας δούμε τώρα πόσο αποτελεσματικά αντιμετωπίζεται η διαφθορά από τα κράτη-μέλη. Η ε, ομολογεί ότι σήμερα δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός να ελέγχει και να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των μέτρων κατά της διαφθορά σε κοινοτικό, σε ενωσιακό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο έχουμε μόνο το Συμβούλιο της Ευρώπης, αλλά και εκεί ε, αυτό το μηχανισμό Συμβούλιο της Ευρώπης που λέγεται Γκρέκο δεν είναι ιδιαίτερα ορατός ε, στα κράτη-μέλη. Επίσης από τον ΟΣΑ που έχει μία σύμβαση για την αντιμετώπιση της δωροδοκίας δημοσίων υπαλλήλων σε διεθνείς συναλλαγές. Γνωρίζουμε λοιπόν από τον ΟΣΑ ότι ενεργός δωροδοκία έλαβε χώρα μόνο σε τέσσερα κράτη-μέλη και η σύμβαση αυτή ισχύει σε 12 κράτη-μέλη. Δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς αντιμετωπίζουμε το όλο θέμα ε, με νομικά μέσα, διότι έχουμε, διαθέτουμε πολλά εξ αυτών τόσο σε ε, διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο. Το ερώτημα που βάζω εγώ είναι πώς ακριβώς χρησιμοποιούνται αυτά τα νομικά εργαλεία. Πρώτα απ' όλα λοιπόν ας δούμε πώς ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προστατεύει η ίδια ε, τα οικονομικά της συμφέροντα από την ε, διαφθορά και πώς το πράττει αυτό σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης. Θα σας αναφέρω τις περιπτώσεις της Όλαφ. Νομίζω ο κύριος Ταβάρης είπε ότι η Όλαφ είναι αποτελεσματική. Θα ήθελα να σας διαβάσω κάτι από τον αρμόδιο Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κύριο Σεμέτα και παραθέτω. Από το έτος 2.281 περιπτώσεις από τις 647 που παρέπεμψε η Όλαφ σε εθνικές δικαστικές αρχές απορρίφθηκαν. Άρα οι μισές απορρίφθηκαν. Στις υπόλοιπες μισές το ποσοστό καταδίκης ήταν ανήλθε σε 41%. Άρα δηλαδή στην Ευρώπη όπου έχουμε τα 20 εκατομμύρια μικροδοροδοκίες ανά έτος, εξ αυτών το πολύ πολύ οι 150 να οδήγησαν σε καταδίκη μετά από πρωτοβουλία της Όλαφ και αυτό σε διάστημα 10 ετών. Είναι λοιπόν πολύ πιο εύκολο να αγοράσει κανείς... Ε, είναι λοιπόν πολύ πιο εύκολο να κερδίσει κανείς το λαχείο. Οι πιθανότητες να κερδίσει κανείς λαχείο είναι περισσότερες από το να καταδικαστεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Ας δούμε τώρα τα εργαλεία που υπάρχουν. Υπάρχουν διαφορές στο νομικό πλαίσιο των κρατών μελών και πάλι ε, παραθέτω εδώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν λοιπόν ε, οργανωτικοί φραγμοί σε υπερεθνικές ε, έρευνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό σημαίνει ότι δεν προστατεύονται σωστά στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα συμφέροντα αυτής. Και η ίδια η Όλαφ λέει έχουμε 300 ε, περίπου ε, περιπτώσεις όπου μας δίδονται πληροφορίες ανέτος. Επειδή όμως λέει ένας διευθυντής όλευ δεν έχω ε, αρκετό προσωπικό, δεν μπορώ να εξετάσω όλες αυτές τις περιπτώσεις. Η ίδια η Όλαφ ομολογεί ότι δεν έχει λοιπόν αυτό το δυναμικό. Ο διευθυντής ο ίδιος τον οποίο παραθέτω, τα λόγια του οποίου παραθέτω, λέει ότι εγώ δεν μπορώ να ψάξω μόνος μου τον τραπεζικό λογαριασμό των υπόπτων. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα, ότι η Όλαφ ε, δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλία για έρευνες, απλά έρευνα μετά από αναφορά πληροφοριών. Άρα λέει τα καταφέρει κανείς, αν τα καταφέρνει κανείς ε, στον τομέα του να παραμείνουν όλα τα στόματα κλειστά, ε, δεν γίνεται καμία έρευνα. Τελειώνει και η ιστορία, γιατί η Όλαφ δεν έχει ούτε το προσωπικό, ούτε τις αρμοδιότητες να λειτουργήσει αποτελεσματικά, διότι δεν μπορεί καν, δεν έχει το δικαίωμα να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να το ετηθεί μέσω τρίτων. Η Κομισιόν λοιπόν άρχισε να δουλεύει αρκετά σοβαρά για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Όμως ε, εξακολουθούμε να βρισκόμαστε στα πολύ πρώτα στάδια. Για πρώτη φορά υπάρχει ε, έκθεση κατά της ε, διαφθοράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η έκθεση από το 2013 και εφεξής θα αρχίσει να δημοσιεύεται ανά δύο έτη. Η, Ευρωπαϊκή, η Κομισιόν τον Ιούνιο ε, προτίθεται να καταθέσει μία πρόταση για το αξίωμα του δημόσιου κατήγορου και έχει ήδη ξεκινήσει με προτείνοντας ε, μια συγκεκριμένη οδηγία για την εναρμόνιση του ποινικού δικαίου στα κράτη-μέλη από το 2013 και εφ' και επίσης έχει καταθέσει και πρόταση για μεταρρύθμιση της Eurojust και αυτό από το 2013 και μετά. Άρα δηλαδή βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, λαμβάνει ορισμένα σημαντικά μέτρα. Παρόλα αυτά, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενθάρρυνση από το Κοινοβούλιο. Τώρα, τι κάνουν ακριβώς τα κρατη Όχι και πολλά. Θα σας ε, αναφέρω μόνο μία περίπτωση για να κατανοήσετε το συλλογισμό μου. Ακόμα λοιπόν και σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται διαφθορά αλλοδαπών υπαλλήλων, αυτό σε πολλές περιπτώσεις σημαίνει δωροδοκία σε κυβερνήσεις ε, άλλου κράτους μέλους. Και αυτό έχει συμβεί. Η αντίδραση του κράτους μέλους, του κράτους του συγκεκριμένου, ήταν πολύ φτωχή σε ένα κράτος μέλος υπήρξαν αντιδράσεις σε πάρα πολλά άλλα κλείνει το θέμα. Παρότι τα κράτη αυτά έχουν υπογράψει, όπως σας είπα, την σχετική συμφωνία του ΟΣΑ. Πάντως τα αποτελέσματα, μιλάμε τώρα για ένα μεγάλο κρατοσμέλος, ήταν τα εξή. Από το 2005 και εφ' εξή, και αυτά τα στοιχεία προέρχονται από την έκθεση του ΟΣΑ. Από το 2005 μέχρι το τέλος του 2010, 69 άτομα ε, καταδικάστηκαν, εκ των οποίων 30 ε, καταδικάστηκαν σε ποινικό επίπεδο και οι υπόλοιποι ε, απλά επέστησαν οικονομικές κυρώσεις τους. Επιβλήθηκαν ε, πρόστιμα και μάλιστα το όνομά τους δεν έγινε καν γνωστό ε, στην κοινή γνώμη. Από τους 30 ε, μερικοί καταδικάστηκαν με αναστολή και μόνο τέσσερις πραγματικά εγκλίστηκαν σε σοφρονιστικά καταστήματα. Και επίσης πάλι τέσσερις καταδικάστηκαν για σοβαρές υποθέσεις, για, μιλάμε τώρα για εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Άρα δηλαδή, ακόμα υπολείπονται πάρα πολλά ε, σε επίπεδο κρατών μελών και στα κρατη υπάρχουν περιπτώσεις ε, όπου ολόκληροι τομείς πλήττονται από συστημική διαφθορά. Και αυτά τα στοιχεία έρχονται από την ε, Transparency International. Ε, κράτη λοιπόν όπου εμπλέκονται οι δημόσιοι υπάλληλοι και είναι δύσκολο ακόμα και για τους πολίτες να αντιδράσουν σε αυτά τα κρατημέλη, να αντιδράσουν κατά αυτού του φαινομένου. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα και πάρα πολλοί από εμάς δεν θα θέλαμε ούτε καν να τη γνωρίζουμε. Τελειώνοντας λοιπόν θα ήθελα να ε, προβώ μένες γενικής φύσεως παρατηρήσεις. Και σε συγκεκριμένα σχόλια. Στι Ηνωμένε Πολιτείες κατά τα τέλη του 19ου αιώνα εμφανίστηκε το προοδευτικό κίνημα το οποίο συνέστησε ισχυρούς ομοσπονδιακούς ε, θεσμούς για να αντιμετωπιστεί η ευρέως διαδεδομένη διαφθορά τότε στις ΗΠΑ. Ε, FBI, IRS, νομίζω λοιπόν ότι χρειαζόμαστε ε, κάτι πιο ισχυρό, όχι απλά τον δημόσιο κατήγορο, τον ΕΠΟ όπως λέγεται, τον εισαγγελέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να υπάρχει μια πιο ισχυρή ευρωπαϊκή αρχή έτσι ώστε να μπορέσει να σπάσει τον φαύλο κύκλο της συστημικής διαφθοράς σε πολλούς τομείς και σε πολλά κράτη-μέλη. Οι φορολογούμενοι ε, επιθυμούν να χρησιμοποιούμε σωστά τα χρήματά τους, κυρίως στο Βορρά, αλλά ακόμα και στο Νότο. Οι φορολογούμενοι επιθυμούν να είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί και νομίζω μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό. Ε, με συγχωρείτε που μακρηγόρησα γιατί ξέρετε ε, έχω παθιαστεί με το θέμα αυτό. Έχω βέβαια και συγκεκριμένες προτάσεις, μπορείτε να τις διαβάσετε. Αυτό όμως που θέλω να κρατήσετε από την ομιλία μου είναι όχι οι προτάσεις, αλλά εκείνο που μέχρι τώρα έχουμε παραβλέψει. Ευχαριστούμε κύριε Σκυλακάκη και θα έχουμε χρόνο και για τις λεπτομεριακές προτάσεις. Είπα ότι η Όλαφ έχει σημαντικές εξουσίες. Τώρα το κατά πόσο τις χρησιμοποιεί αποτελεσματικά ή όχι, νομίζω ότι ήταν πολύ βάσιμο και το δικό σας επιχείρημα προς την άλλη πλευρά ίσως, αλλά δεν θα ήθελα τώρα να επισέλθουμε σε αυτή τη συζήτηση. Ας ολοκληρώσουμε την παρουσίαση των θεματικών εγγράφων, δίνοντας το λόγο στον κύριο Ντεγιόγκ, που θα μιλήσει για τη διαφθορά σε ιδιωτικέ επιχειρήσει που διαταράσσουν το θεμητό ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Ο κύριος Δεγιόνγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα δύο εισαγωγικέ παρατηρήσεις να υποβάλω. Καταρχήν, ε, θα διαπιστώσετε, το δικό μου έγγραφο είναι πολύ πιο σύντομο από τα προηγούμενα, <laughs> γιατί τήρησα, εγώ τήρησα τα τυπικά κριτήρια και τα τυπικά όρια που μας επιβάλλονται. Ε, βέβαια, διαπίστωσα ότι τελικά δεν ήταν τόσο αυστηρά τα κριτήρια αυτά όσο φαινόταν. Θα μπορούσα να είχα υποβάλει πολύ περισσότερα στατιστικά και αριθμητικά στοιχεία. Υπάρχουν αρκετές συστάσεις ε, στο εγγραφό μου, αλλά η εισαγωγή και κυρίως η παρουσίαση του προβλήματος είναι αρκετά συνοπτική εξαιτία ε, του περιορισμού που έχουμε από τις σελίδες, ε, ε, στις σελίδες των εγγράφων. Κύριε Σκυλακάκη, πολλά από αυτά που είπατε εσείς ε, θα μπορούσαν να είχαν περιληφθεί στο δικό μου έγγραφο. Άρα τέλος καλό, όλα καλά. Αν συνδυάσετε τα στατιστικά αριθμητικά στοιχεία που μας παρουσίασε ο κύριος Σκυλακάκης και τα συμπεράσματα του δικού μου εγγράφου θα διαμορφώσετε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το θέμα αυτό. Το θεματικό μου έγγραφο επίσης αντανακλά την προσπάθεια που έκανα και στην ε, Επιτροπή Ιστορικής Αγοράς ε, να ε, αναγάγω αυτό το θέμα σε σημαντική προτεραιότητα προκειμένου να περιληφθεί και σε μια έκθεση πρωτοβουλίας. Όπως φάνηκε από τη σύντηση των συντονιστών, τελικά προτιμήθηκε αυτό το θέμα στη δική μας Επιτροπή από ό,τι στην Επιτροπή Ιστορικής Αγοράς. Αλλά το θέμα αυτό αφορά και την Επιτροπή Ιστορικής Αγοράς γιατί θέλουμε να εξασφαλίσουμε όντως θήκες θεμητού ανταγωνισμού στην ε, ενιαία, στην εσωτερική αγορά. Και νομίζω ότι είναι λέδα αυτά τα θέματα, γιατί εφόσον οι επιχειρήσεις ε, ε, δωροδοκούν αλλοδαπού δημοσίου λειτουργού, όχι στου ημεδαπού, και δεν διώκονται, τότε το κλίμα για τις επιχειρήσεις ε, είναι πολύ πιο ελκυστικό και πρόσφορο στις ε, χώρες που βρίσκουν λειτουργούς να δωροδοκίσουν. Είναι αλληλένδετα λοιπόν αυτά τα θέματα διαφθοράς και θεμητού ανταγωνισμού και σίγουρα επηρεάζουν τον ανταγωνισμό και τις συνθήκες θεμητού ανταγωνισμού στην εσωτερική μας αγορά. Δεύτερη παρατήρηση. Αν διαβάσετε και την έκθεση της κυρίας Γκάμπριελ για τις δημόσιες προμήθειες και εκεί φαίνεται πόσο στενά άρρηκτα συνδεδεμένη είναι η εσωτερική αγορά και το θέμα των δημοσίων προμηθειών και υπάρχει σχετική οδηγία με το θέμα της διαφθοράς και επηρεάζεται αυτό το θέμα και επηρεάζει αυτό το θέμα και τις δικές μας εργασίες. Γι' αυτό και πιστεύω θα πρέπει να έχουμε στενή συνεργασία με την Επιτροπή Εσωτερική Αγοράς. Αν δείτε τα αποτελέσματα στην ε, εφαρμογή, πραγματικά με σόκαρε η 8η έκθεση, της έκθεση πρόοδου για την εφαρμογή της ε, συνθήκης του ΩΣΑ που αφορά τη δωροδοκία των αλλοδαπών δημοσίου λειτουργών. Είναι μια πολύ ειδική συνθήκη του ΩΣΑ αφορά ακριβώς αυτό το θέμα. Είναι πολύ εύκολη, σύντομη, ε, συγκεκριμένη και πολύ σημαντική η συνθήκη αυτή του ΩΣΑ και μάλιστα θεσπίστηκε μια εποχή που μόνο οι ΙΠΑ είχαν σχετική νομοθεσία που ποινικοποιούσε τη δωροδοκία των, δημοσίων, των αρδαπών δημοσίων λειτουργών. Και ε, με ένα τέτοιο νομοθέτημα δημιουργόταν και παγκοσμίω πιο ε, ε, θεμητές συνθήκες ανταγωνισμού. Και αυτό συνέβη με τη συνθήκη του ΟΣΑ, γιατί υπήρχε μια ε, διαδικασία ε, εκτέλεσης και εποπτείας με βάση τον έλεγχο ομοτήμων. Είναι πάντως αξιοσημείωτο που ακόμη και μέχρι σήμερα πέντε χώρες μέλη δεν έχουν ακόμη κυρώσει τη συνθήκη αυτή του ΟΣΑ. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή, αυτή η ετήσια έκθεση κατέληξε το συμπέρασμα ότι 11 α, χώρες είχαν ε, ίσονο α, περιπτώσεις διώξεων, ε, τέσσερις είχαν πάνω από τρεις α, σημαντικές περιπτώσεις διώξεων και μερικές χώρες δεν είχαν καν ξεκινήσει καμία δίωξη για τέτοια θέματα. Και αυτό εξηγείται εν μέρει από το γεγονό ότι μερικές χώρες μέλη έχουν περισσότερε εταιρείε με διεθνεί δραστηριότητες από άλλε. Η δική μου πατρίδα, 100 χώρε, για παράδειγμα, Δυστυχώ έχει ε, ελάχιστη, ε, πολύ κακέ επιδόσει ό,τι αφορά την εφαρμογή τη συνθήκη του ΩΣΑ. Δεν υπάρχει καμία, δίκη και κατα... δεν υπάρχει καμία καταδίκη και ελάχιστε ε, έρευνε και ανακρίσει γίνονται. Παρόλο που η Ολλανδία αποτελεί την έδρα πολλών πολυεθνικών εταιριών. Και μάλιστα και το φορολογικό μας περιβάλλον ενθαρρύνει την εγκατάσταση πολυεθνικών εταιριών στην Ολλανδία. Άρα κάτι δεν πάει καλά. Κάτι πάει στραβά. Δεν υπάρχει. Δεν πιστεύω ότι δεν μπορεί ο, ο δημόσιος κατήγορος ε, δεν έχει τη, τη συγκεκριμένη τεχνογνωσία. Βέβαια είναι περίπλοκες αυτές οι περιπτώσεις ε, για την εισαγγελία είναι δύσκολο να συγκεντρωθούν αποδεικτικά στοιχεία και άμα είναι και διασυνοριακή υπόθεση, η συλλογή αποδείξεων και γενικώ η δίωξη γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη. Αλλά είναι και τεράστια τα συμφέροντα στην εσωτερική αγορά. Γι' αυτό και πιστεύω ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να μας απασχολήσει. Και αυτό είναι, αυτή είναι η πρώτη μου σύσταση. Θα πρέπει να εξασφαλιστούν συνθήκε θεμητού ανταγωνισμού και αυτό θα γίνει με την κύρωση και εφαρμογή από όλα τα κράτη-μέλη των διεθνών συμβάσεων του ΟΗΕ, του ΟΣΑ για την πάταξη της ε, δωροδοκίας. Αυτή είναι μια σημαντική βάση και σε ό,τι αφορά την εφαρμογή θα πρέπει να γίνει συζήτηση μεταξύ των κρατών μελών για το πώς θα εκτελεστούν, πώς θα εφαρμοστούν και εμπράκτως αυτές οι συνθήκες και συμβάσεις οι διεθνείς. Γιατί υπάρχουν μεγάλες διαφορές όπως σας είπα. Ε, οι επιδόσεις της ε, Ολλανδίας είναι πολύ κακές. Το Ηνωμένο Βασίλειο προσπαθεί να αφιερώσει πολύ περισσότερους πόρου στο θέμα αυτό και μακάρι θα ήταν πολύ γόνιμο, πιστεύω, να γίνει συζήτηση και μεταξύ αυτών των δύο χωρών, αλλά και μεταξύ των 27 χωρών μελών, για να δούμε τι εμπειρογνωμοσύνη χρειάζονται, πόσο αποτελεσματικέ είναι ε, οι υπηρεσίε που ασχολούνται με την εφαρμογή, πόσο συνεργάζονται και αν μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα ελάχιστο ποσοστό πόρων που θα πρέπει να αφιερώνουμε στο θέμα αυτό. Οι δεμή θα συνεχιστούν αυτές οι μεγάλες διαφορές εφαρμογής μεταξύ των κρατών μελών. Γι' αυτό και προτείνω να καταλήξουμε σε, κάποια, σε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των συνθήκων αυτών και φυσικά να χρησιμοποιηθεί το δίκτυο των σημείων επαφής ε, που υπάρχουν για τη διαφθορά σε όλα τα κράτη-μέλη. Γιατί κάθε χώρα έχει ορίσει έναν αξιωματούχο ειδικό, ένα σημείο επαφής ε, για θέματα πάταξης της διαφθοράς. Και συνήθως αυτά τα σημεία επαφής βρίσκονται στη, στις Οπότε θα πρέπει τα σημεία επαφή να γίνουν πιο αποτελεσματικά στο έργο του αυτοί οι αξιωματούχοι, γιατί φαίνεται ότι βρίσκονται σε λανθάνουσα ακόμη κατάσταση αυτοί οι φορεί. Δεν φαίνεται να λειτουργούν, γιατί έχουμε ένα δίκτυο, γιατί να μην το αξιοποιούμε. Μπορούμε να ανταλλάσσουμε τις βέλτιστες πρακτικέ και να εκπονούμε τι κατευθυντήριε γραμμέ που θα εφαρμόσουν στη συνέχεια τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν όμω και κάποια νομικά θέματα που θα πρέπει να διευκρινιστούν. Και εκεί ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να αναλάβει κάποια πρωτοβουλία. Το θέμα τη ε, ποινική ευθύνη των νομικών προσώπων, για παράδειγμα, είναι ένα οριζόντιο θέμα στο ποινικό δίκαιο. Γιατί δεν το γνωρίζουν αυτό όλα τα κράτη-μέλη. Είναι σημαντικό το θέμα. Γιατί αν μόνο, φυσι... ιδιώτε, φυσικά πρόσωπα μπορούν να διώκονται, τότε περιορίζουν... περιορίζεται η αποτελεσματικότητα του ποινικού δικαίου σε ό,τι αφορά την πάταξη τη διαφθορά. Ένα δεύτερο νομικό πρόβλημα που δημιουργεί τεράστιο ε, δυσκολία στα κράτη-μέλη είναι η ευθύνη στις μητρική εταιρεία για τις θυγατρικές της εταιρείες. Είχαμε μια πολυνική υπόθεση όπου θυγατρικές της ε, Philips ε, μέτρα την Ολλανδία καταδικάστηκαν για δωροδοκία νοσοκομιακού προσωπικού είναι δημόσιοι λειτουργοί και οι Ολλανδοί δεν έλαβαν κανένα μέτρο, καμία δίωξη δεν έκαναν κατά τη Φίλιψη γιατί θεώρησαν ότι η Φίλιψη η μητρική δεν μπορεί να ευθύνεται για τι θηγατρικέ τη στην Πολωνία. Υπάρχει λοιπόν έλλειψη ασφάλεια δικαίου ω προς τις σχέσεις μεταξύ μητρικής και θηγατρικών εταιριών, κάτι που δυσκολεύει την διαλεύκανση των υποθέσεων. Και ένα άλλο θέμα που είναι πολύ γνωστό όσοι ασχολούνται με τη συνθήκη του ΩΣΑ και εξετάζεται πολύ, πολλά χρόνια το θέμα το facilitation of payments, τη πληρωμέ της πληρωμές διευκόλυνσης που κατά κάποιο τρόπο τις επιτρέπει ε, η συνθήκη του ΩΣΑ. Δηλαδή, αν έχει κανείς κάποια αγαθά και περιμένουν στα λιμάνια, μπορεί να καταβάλει ένα μικρό ποσό για να ε, θεωρηθούν ως προτεραιότητα. Αυτό μπορεί να, να θεωρηθεί ως πληρωμή διευκόλυνσης Βέβαια, ο ορισμός είναι κάπως ασαφής, απροσδιόριστος ε, και γενικώ ε, όταν μιλάμε με κράτη-μέλη και μη κυβερνητικέ οργανώσεις λένε ότι θα πρέπει είτε να βελτιωθεί ο ορισμός είτε να καταργηθεί τελείως αυτό το θέμα των πληρωμών διευκόλυσης γιατί είναι πολύ ρευστά τα όρια μεταξύ του τι εστία τέτοια πληρωμή διευκόλυσης και τι εστί δωροδοκία. Θα μπορούσε λοιπόν για όλα αυτά τα θέματα να υποβάλει προτάσεις για τη διαλεύκαση του νομικού πλαισίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να το συζητήσουμε κι εμείς. Πέρυσι είχαμε πολύ γόνιμο διάλογο με τον επιτρόπο Μάμστρομ και εδώ παρουσιάστηκε το σχέδιο δράση κατά της διαφθοράς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλιστα ήταν πολύ θετική η ανταπόκριση της Επιτρόπου. Βέβαια, υπάρχουν κάποιε διαφορέ ω προ την γενική προσέγγιση. Αντιλαμβάνομαι ότι του χρόνου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει μια εμπεριστατωμένη έκθεση. Αλλά τι γίνεται στο μεταξύ, δεν θα υποβληθούν νέε νομικέ ε, προτα... νομοθετικέ προτάσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί έτσι θα χαθεί πολύτιμο χρόνο. Και για τι δημόσιε προμήθειε, ειδικά, θα μπορούσαμε παράλληλα να είχαμε κάποιε πρωτοβουλίε για να εφαρμόσουμε καλύτερα την νομοθεσία κατά τη διαφθοράς που επηρεάζει τι δημόσιε προμήθειες. Και αναφέρθηκα σε τρεις τομεί που χρήζουν διευκρίνηση. Κατά τη γνώμη δεν χρειάζεται να περιμένουμε την επόμενη έκθεση για να, για να υποβληθούν και πρωτοβουλίε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη να αναλάβει νομοθετικέ πρωτοβουλίε στο θέμα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρί να περιμένει τη δημοσίευση τη επόμενη έκθεση. Αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να βελτιώσει τη μεθοδολογία του. Γιατί κάθε χρόνο έχουμε εκθέσει από τον ΟΣΑ, από τον Γκρέκο, από το Συμβούλιο τη Ευρώπη. Αλλά δεν υπάρχει διαρθρωμένο τρόπο αντιμετώπιση και εξέταση αυτών των εκθέσεων. Πιστεύω ότι αξίζουν οι εκθέσει αυτέ προσοχή και συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί αναλύει την κατάσταση στα κράτη-μέλη είναι αντικείμενο διαπραγματεύσεων και οι συστάσεις του ΩΣΑ και οι συστάσεις του Γκρέκο. Και από εκεί έχουμε να αντλήσουμε πάρα πολλά διδάγματα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα αυτό το υλικό ως βάση για το δικό μας έργο. Πέραν της έκθεσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιστεύω ότι έτσι θα εμπλουτιστεί πολύ περισσότερο η συζήτησή μας. Αυτά προς το παρόν νομίζω ότι οι συστάσεις μου μιλάνε από μόνος τους. Μπορούμε να περάσουμε στη συζήτηση τώρα. Ευχαριστούμε κύριε Ντεγιόγκ. Έχουμε διαμορφώσει πια μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις τέσσερις ε, θεματικές ενότητες, δημόσιες προμήθειες, ε, κοινοτικά κονδύλια, συστημική διαφθορά στις δημόσιες διοικήσεις και έλλειψη ε, θεμητού ανταγωνισμού εξαιτία τη διαφθορά μεταξύ των επιχειρήσεων στην εσωτερική αγορά. Αυτέ ήταν οι τέσσερι θεματικέ ενότητε, τα τέσσερα έγγραφα και γίνονται και πολύ σημαντικέ συστάσει προ τα θεσμικά όργανα. Θα έχουμε τώρα συζήτηση, θα λάβουν τώρα πρώτα το λόγο οι συντονιστέ, όσοι συντονιστέ είναι παρόντε από τι πολιτικέ ομάδε. Θα ακούσουμε κατόπιν του ευρωβουλευτέ και μετά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναρωτιέμαι να έχουμε εκπρόσωπο και του Συμβουλίου. Όχι, μόνο η Επιτροπή θα λάβει το λόγο. Οπότε με, θα μπορούσε και τις δικές μας θέσεις να τις διαβάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη-μέλη, κυρίως την ανάγκη να κυρωθούν το συντομότερο δυνατό οι συνθήκες του ΟΗΕ και του ΟΣΑ από τα κράτη-μέλη που έχουν ολιγορήσει το θέμα αυτό. Άλλωστε αυτό το προτείνουν και οι εισηγητές μας. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι δυνατότητε έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως νομικό πρόσωπο να συνυπογράψει το μέλλον διεθνείς συνθήκες και υπάρχει πιθανότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσχωρήσει σε τέτοιου είδου συνθήκες για την πάταξη της διαφθοράς. Αυτά. Περνάμε στη συζήτηση λοιπόν. Πρώτα οι συντονιστέ και μετά οι υπόλοιποι ευρωβουλευτέ. Θα ξεκινήσουμε από την κυρία Ματιού που εκπροσωπεί το ΕΛΚ. Λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τους ε, τέσσερις ε, ομιλητές ε, που παρουσίασαν τις θεματικές αυτές και που πραγματικά μας διευκρίνησαν με πολύ ενδιαφέροντο τρόπο ο καθένας στον τομέα του. Θεωρώ ότι ήταν, μας εμπλούτησε ιδιαίτερως αυτή, αυτές οι παρουσιάσεις και χαίρομαι πάρα πολύ που θα συμπεριληφθούν στην αναφορά της Επιτροπής μας, στην έκθεση της Επιτροπής μας. Θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό αυτό. Μας δίνουν τέσσερις οπτικές γωνίες και μας δίνουν κάποιες βάσεις εργασίας για να ε, προσπαθήσουμε να πατάξουμε τη διαφθορά. Και οι τέσσερι παρουσίε βεβαίω μα είπαν ότι είναι δύσκολο να έχουμε συγκεκριμένα νούμερα όσον αφορά τι ζημίε που προκαλεί η διαφθορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά όσον αφορά τα ενδιαφέροντα στοιχεία, ε, μας είπε η κυρία Γκαμπριέλ ότι αυτό το οποίο είναι ιδιαίτερο επιζήμιο είναι η έλλειψη της ε, εφαρμογής των οδηγιών σε ορισμένες χώρες μέλη και θεωρώ ότι θα έπρεπε να προσπαθήσουν γιατί είναι εδώ και 8 χρόνια που θα έπρεπε να μεταφέρουν αυτές τις οδηγίες σε εθνικό επίπεδο και Νομίζω ότι πραγματικά θα έπρεπε να κάνουμε μια προσπάθεια μεταφοράς της ε, οδηγίας. Γιατί αν δεν γίνει αυτό δεν θα μπορέσουμε να πατάξουμε αποτελεσματικά τη διαφθορά και να έχουμε ορισμένα αποτελεσματικά εργαλεία που να σε επιτρέψουν μια καλύτερη προσέγγιση του φαινομένου αυτού. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να ε, επισπεύσουμε τις προσπάθειές μας για την ε, μεταφορά αυτή των οδηγιών σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, όσον αφορά τη σύναψη με τις συμφωνίες με τον ΟΣΑ, και οι τέσσερις ομιλητές έθιξαν το θέμα αυτό και εδώ υπάρχουν κάποιοι, κάποιες χώρες μέλη που είναι, δείχνουν ε, ότι είναι κακοί μαθητές και νομίζω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε υπό την ιδιότητά μας ως βουλευτών να στις κυβερνήσεις υπογράψουν αυτές τις συμφωνίες του ΩΣΑ θα αναμένουμε βεβαίω τη θέση τη Επιτροπή όσον αφορά τη δημιουργία τη ίστα Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γίνεται ευρέω ε, λόγο για το θέμα αυτό στο ιστορικό των πολιτικών ομάδων και ελπίζω ότι, εν πάση περιπτώσει, ε, θα δούμε ποια θα είναι βεβαίω η πρόταση τη Επιτροπή. Ε, και εγώ πραγματικά την αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί ελπίζω ότι αυτοί οι νομικοί θα έχουν μια θετική επίπτωση όσον αφορά την αποτελεσματική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Εκτίμησα ιδιαίτερο τα είπε ο κ. Σκυλακάκης για την Όλαφ και με κατέπληξε ε, ο πολύ μικρός αριθμός από καταδίκες στην Όλαφ, γιατί γνωρίζουμε ότι η Όλαφ εργάζεται σοβαρά, διεξάγει πολλές έρευνες, όσο δεν είναι παρκής, δεν είναι αρκετές. Ε, Αισθάνθηκε κάποια απογοήτευση όταν μας μιλήσετε για τα πολύ πενιχρά αποτελέσματα τελικά. Ίσως θα μπορέσουμε να μιλήσουμε σχετικά με το θέμα αυτό σε ένα άλλο πλαίσιο ή αργότερα. Ε, Συγχαρητήρια λοιπόν και πάλι προς, και, προς τους τέσσερις ομιλητές. Α, και κάτι άλλο όσον αφορά την ενίσχυση της πληροφόρησης των ε, αστυνομικών αρχών. Ε, μιλούμε για το θέμα αυτό στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και όταν ε, ακούμε τι γίνεται στη ΣΕΠΟΛ νομίζω δεν δικαιολογείται η συγχώνευση μεταξύ ΣΕΠΟΛ και Europol. Νομίζω ότι στη ΣΕΠΟΛ, η ΣΕΠΟΛ θα πρέπει να υποστηριχθεί για μια πραγματικά καλύτερη κατάρτιση των αστυνομικών αλλά και των ε, νομικών, ε, των δικαστικών λειτουργών. Και ε, νομίζω ότι θα μπορούσαν και αυτοί να έχουν μια καλύτερη κατάρτιση όσον αφορά την πάταξη διαφθοράς δικαστική. Ε, αλλά θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να διατηρηθεί η ΣΕΠΟΛ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ματιέ. Τώρα θα περάσουμε, ε, θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Φαγιόν ε, για τους εκ σοσιαλιστών. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τους ε, συναδέλφους ε, και τους τέσσερις γιατί έκαναν πραγματικά μια πολύ καλή δουλειά. Νομίζω ότι όλα αυτά αποτελούν μια πολύ καλή βάση για τη σημερινή συζήτηση. Πιστεύω ότι ο εισηγητής μας, ο κύριος Γιακολίνο, ε, θα τα μελετήσει όλα αυτά σε βάθος ε, και θα είναι πολύ καλά προετοιμασμένος όταν ε, θα καταθέσει την έκθεσή του. Άκουσα σήμερα να γίνεται λόγος για πολλά πορίσματα και κατέληξα στο συμπέρασμα ε, στο ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν τα καταφέρνουμε και πολύ καλά στο να αντιμετωπίσουμε τη διαφθορά. Εξάλλου ε, τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους. Κάθε χρόνο χάνουμε από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό 2 δις ευρώ λόγω της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Ας δούμε τώρα τι είναι η διαφθορά. Υπάρχει άραγε κοινός ορισμός της ε, διαφθοράς Μπορούμε να ε, μιλάμε για το πώς μετριέται η διαφθορά, γιατί η διαφθορά έχει σχέση με δύο πλευρές, ε, με την δωροδοκία και την δωροληψία. Ε, μπορούμε λοιπόν να καταλήξουμε σε έναν κοινό ορισμό της διαφθοράς για να μπορούμε πάνω σε αυτό να την αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν πολλές μελέτες που καταδεικνύουν πολλά προβλήματα στην αντιμετώπιση της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα. Ίσως να έχουμε πρόβλημα με τη διαφθορά, διότι δεν είμαστε σε θέση να μετρήσουμε την έκταση της ε, διαφθοράς. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε εμείς ε, με τη μορφή συστάσεων. Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν δομές ε, οι οποίες θα μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε δικαστικά, να καταδικάζουμε όλους εκείνους που εμπλέκονται σε υποθέσεις σε διαφθορά στα κρατη ε, όπου η διαφθορά έχει άμεση ή έμεση σχέση με το οργανωμένο έγκλημα. Βλέπουμε ε, πολλές απάτες στον τομέα του ΦΠΑ και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα ε, που πρέπει να εξετάσουμε γιατί σε αυτό το επίπεδο χάνουμε πολλά χρήματα από το ΦΠΑ. Κάτι άλλο σημαντικό πώς συνεργάζονται μεταξύ τους τα κράτη-μέλη. Σήμερα εξετάζουμε κυρίως τη διμερή συνεργασία. Αλλά τι γίνεται με την πολυμερή. Πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με την Όλαφ ε, είναι επιτυχής η Όλαφ και οποτεδήποτε καταθέτει έκθεση η Όλαφ πώς ανταποκρίνονται στα κράτη-μέλη πώς μετράμε την ε, ε, εφαρμογή των συστάσεων και τι είδους ε, σχόλια προκύπτουν από τις, ε, στις εκθέσεις της Όλαφ. Συμφωνώ με αυτό που είπε η κυρία Ματιού, ότι και η Europol και η ΣΕΠΟΛ είναι σημαντικοί οργανισμοί. Πράγματι, αυτοί οι δύο θεσμοί ε, δεν θα πρέπει να συγχωνευτούν υπό την αιγίδα της Europol. Η Europol αποκτά πολλές αρμοδιότητες σε καθημερινή βάση. Εάν λοιπόν ε, τις παραδώσουμε και την ΣΕΠΟΛ, τα πράγματα θα γίνουν πολύ πιο δύσκολα. Να γίνουν περισσότερα στην ε, κατάρτιση, την εκπαίδευση όλων εκείνων που ε, καταπολεμούν τη διαφθορά. Ακούσαμε πολλά σχόλια για το ε, αξίωμα του Ευρωπαίου Ισαγγελέα. να συσταθεί αυτό το αξίωμα. Πιστεύουμε ότι αυτή είναι μια ιδέα που πρέπει να προχωρήσει με πολύ σύνεση να δούμε τι είδου ε, θεσμοί είναι χρήσιμοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πάντως, πρέπει να ε, εκδώσουμε εντολή για το ε, γραφείο, το αξίωμα αυτό του εισαγγελέα που όπως σας είπα θα μπορέσει να καταπολεμήσει τη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα. Ευχαριστώ και πάλι τους ε, συντάκτες και τους τέσσερις αυτών των υποθεμάτων γιατί αυτά που μας είπαν αποτελούν μια πολύ καλή βάση για τη μελλοντική μας δουλειά. Ε, υπάρχουν λοιπόν πολλές αναλύσεις επί του θέματος. Ε, την Τετάρτη θα συζητήσουμε για τη διαφθορά σε εθνικό επίπεδο και νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, περιμένουν από εμά χειροπιαστές συστάσεις. Βεβαίως ε, πρέπει να ασκήσουμε πίεση στις κυβερνήσεις μας για να αναλάβουν ενέργειες. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Ε, μιλήστε πάνω από δύο λεπτά και δεν σας διακόψω γιατί δεν θέλει και κανείς άλλος το λόγο αλλά αν τον θέλετε παρακαλώ γιατί έχουμε ακόμα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον συντονιστή της Άλντε, τον κύριο Νιούτον Ντάν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτές οι τέσσερις συγχύσεις ήταν πραγματικά εντυπωσιακέ. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον παρακαθήμενο συνάδελφο για τις λεπτομέρειες. Ε, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπε και πραγματικά ελπίζω στην τελική μας έκθεση να συμπεριλάβουμε όλες τις συστάσεις των συναντέλφων γιατί σε τελική ανάλυση πρόκειται για ουσιαστικές συστάσεις που θα επηρεάσουν την κοινή γνώμη, τον τύπο, τα κρατημέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εντυπωσιακότατες οι εκθέσεις και συμφωνώ απόλυτα ε, με αυτά που είπε η Τάνια. Ε, λυπάμαι που δεν είναι εδώ ο κύριος Γιακολίνο για να λάβει υπόψη του όλα αυτά που ελέγχθησαν. Ε, κατανοώ βέβαια ότι δεν είναι εδώ η πρόεδρός μας γιατί μου είπε ότι υπάρχει σήμερα, είναι στο, στα δικαστήρια, υπάρχει, εκδικάζεται μια δική της υπόθεση σε σχέση με τη δολοφονία του πατέρα της από τη μαφία. Έπρεπε λοιπόν, έχει, είχε πράγματι αποχρόντα λόγο. Ε, το, κυρία Κάμπρελ, αυτή η κόκκινη ε, σημαία, ε, δεν ξέρω, ε, μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς ακριβώς θα λειτουργούσε αυτό το σύστημα, γιατί εγώ είμαι ποδοσφαιρόφιλο και ξέρω μόνο την κόκκινη κάρτα. Την κόκκινη σημαία δεν την γνωρίζω. Ε, μετά, ε, στην επόμενη μιλήτρια, το θέμα, η κυρία Βάιλερ δεν είπε ακριβώς ε, πώς χρησιμοποιεί η μαφία τα κονδύλια. Μήπως ξέρει που κατευθύνονται, που διοχετεύονται αυτά τα κονδύλια. Ε, την προηγούμενη εβδομάδα ακούσαμε ας πούμε για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Δεν ξέρω πως έχει να μας πει κάτι παραπάνω. Ε, στον κύριο Ντεγιόν, πράγματι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είπατε ε, καλά λόγια για το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά αν το Ηνωμένο Βασίλειο κάνει κάτι, Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει, γιατί ο κύριος Κάμερον είπε να αποσυρθεί το Ηνωμένο Βασίλειο από περιπτώσεις ε, αρρωγής. Ε. Ίσως ε, στο παρελθόν να κάναμε κάτι, δεν ξέρω, για το μέλλον δεν το πολύ βλέπω. Δεν υπάρχει άλλο αίτημα. Θα προσθέσω λοιπόν εγώ ένα δικό μου ερώτημα προς την κυρία Βάιλερ. Ακούμε πολλούς, ε, πολλές για ε, τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προορίζεται τη χρηματοδότηση πολιτικών ε, κομμάτων των χωρών μελών. Μπορείτε να τα επικυρώσετε και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδου φαινόμενα τα οποία γίνονται μέσω ακριβώς συγκεκαλυμμένης χρηματοδότησης είναι, ένα, είναι μια κατηγορία την ακούμε, ε, την ακούμε πολύ συχνά από πολλές χώρες ε, μέλη ε, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το δικό μου ερώτημα. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο και θα δώσουμε το λόγο στον, στην εκπρόσωπο της Κομισιόν, την κυρία Στέφανος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα να παρεύουμε σε αυτή τη ε, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Λέγομαι Τεφενούκ και ασχολούμαι με το φάκελο πάταξη της ε, διαφθοράς την ε, διεύθυνση κομισιών που είναι αρμόδια για αυτό το θέμα, για την πάταξη της διαφθοράς και συνεργάζομαι και με την κυρία Ελισαπέτ Περκινιόν ε, που είναι υπεύθυνη για την ε, καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. μας, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που η κρίμα ασχολείται με το φαινόμενο αυτό γιατί συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των δικών μας προτεραιοτήτων επίσης. Ακούσαμε ε, όλες αυτές τις θεματικές ομιλίες και θεωρήσαμε ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες για το δικό μας έργο που συνεχίζεται. Ε, η Κομισιόν ε, ασχολείται με τον μηχανισμό αναφοράς προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή με τη σύνταξη τακτικών εκθέσεων που βασίζονται σε αξιολογήσεις των χωρών μελών σχέση με τις προσπάθειές τους πάταξης της διαφθοράς. Αυτές οι εκθέσεις θα εκδίδονται κάθε δύο χρόνια και η πρώτη έκθεση θα ε, εκδοθεί, θα παρουσιαστεί ε, στα μέσα του επόμενου έτους και κατά πάσα πιθανότητα θα εγκριθεί το καλοκαίρι, πριν από το καλοκαίρι του 2013. Ε, προσπαθούμε να επικεντρώσουμε στον ε, αντίκτυπο των πολιτικών ε, πάταξη διαφθοράς ε, στο επίπεδο χωρών μελών και στα τελικά αποτελέσματα που έχουμε δει μέχρι τώρα, που έχουμε διαπιστώσει μέχρι τώρα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούσαμε, υπάρχουν εκκλήσεις από την Κομισιόν ε, για να υπάρχουν κάποια επιπρόσθετα όργανα. Εμείς θέλουμε να εστιάσουμε περισσότερο στην πλευρά της εφαρμογής ε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ε, διεθνείς συμβάσεις αλλά λιγοστεί καινούργια νομοθεσία σε αυτό το τομέα. Αυτό το οποίο εμείς επιθυμούμε είναι να επικεντρωθούν οι προσπάθειες στον τομέα της εφαρμογής. Και εμείς εξετάζουμε τόσο αρνητικές όσο και θετικές πρακτικές γιατί το θεωρούμε ότι αυτή είναι μια δεδομένη άσκηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θέσουμε και στις δύο αυτές πτυχές Έχουμε ένα γενικό τμήμα αυτής της έκθεσης, το οποίο θα επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα, το οποίο είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στην πρώτη έκθεση θα εξετάσουμε τη διαφθορά στις δημόσιες προμήθειες συγκεκριμένα και το δεύτερο τμήμα της έκθεσης θα εξετάσει τις ατομικές αξιολογήσεις των χωρών μελών. Έχουμε αξιολογήσει από κάθε χώρα μέλος η οποία εξετάζει αυτό το οποίο θεωρούμε κάποια ιδιαίτερης σημασία ε, θέματα τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη μία την άλλη χώρα. Ε, θέλουμε λοιπόν να εξετάσουμε τις διαμορφίες της κάθε χώρας ε, μέλους, γιατί όπως αναφέρθηκε προηγουμένως υπάρχουν ε, διαφορές όσον αφορά ε, με τις χώρες μέλη, ε, σχέση με αυτό το εκτεταμένο φαινόμενο διαφθορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες, εδώ ακούσαμε μια παρουσίαση πολύ ενδιαφερόντων ε, θεμάτων και στο θέμα αυτό θα επικεντρώσουμε ε, στην πρώτη μας έκθεση που θα εκδοθεί τον επόμενο χρόνο και θα συμπεριλάβει κάποιες ειδικέ συστάσεις. Η Επιτροπή πρότεινε μία αναθεώρηση του νομικού πλαισίου για τις ε, προμήθειες και να έκανε κάποιες προτάσεις για τις δημόσιες προμήθειες ε, που θα αφορούν τις εταιρείε κοινή ωφέλεια και τις παραχωρήσεις δημοσίων έργων. Ε, έχουμε κάνει κάποιες προτάσεις για αρκετές διατάξεις που στοχεύουν στην πολιτική πάταξη διαφθοράς ιδιαίτερα στον τομέα των δημοσίων προμηθειών. Για πρώτη φορά η οδηγία τις, για τις δημόσιες ε, προμήθειες περιλαμβάνει μια διάταξη που αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων και που θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ, σημαντικό θέμα όταν ασχολούμαστε με το θέμα αυτών των δημοσίων προμηθειών και επίσης έχουμε ε, προτείνει ε, ένα σύνολο διατάξεων μεγάλης εμβέλειας όσον αφορά τη λεγόμενη διακυβέρνηση, δηλαδή ένα σύνολο διατάξεων που αφορούν ε, τα θέματα της εποπτείας, κάτι το οποίο αναφέρθηκε επίσης στις θεματικές ομιλίες, επίσης θέματα που σχετίζονται με αυτό το σύστημα συναγερμού, τις κόκκινες σημαίες, που επιτρέπουν στην κάθε χώρα μέλος να ε, αναγνωρίσει, να διαπιστώσει με έναν, από μια κεντρική θέση ορισμένους δείκτες όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες, δείκτες διαφθοράς όσον αφορά τις δημόσιες ε, προμήθειες και θα συμπεριληφθούν όλα αυτά στην αναθεώρηση τη οδηγία για τι δημόσιε προμήθειε. Επίσης υπάρχουν σημαντικές διατάξεις όσον αφορά ζητήματα εποπτείας για μια κεντρική βάση δεδομένων που σχετίζονται με περιπτώσεις διαφθοράς και σύγκρουση συμφερόντων στον τομέα των δημόσιων προμηθειών. Ελπίζουμε ότι θα ακολουθήσει τη συζήτηση θα παρακολουθήσουμε τη συζήτηση όσον αφορά την ε, έγκριση αυτών των ε, διατάξεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, διατάξει όσον αφορά τη χρηστή διακυβέρνηση και τη σύγκρουση οικονομικών συμφερόντων ειδικότερα. Όσον αφορά τα άλλα θέματα που αναφέρθηκαν εδώ, θα πρέπει να πω ότι πράγματι τα θέματα αυτά ε, βρίσκονται στο επίκεντρο του έργου και των προσπαθειών της Επιτροπής για την έκθεση κατά της διαφθοράς όσον αφορά την ατομική ε, αξιολόγηση κάθε χώρας, ε, ασχολούμεθα με την αποτελεσματικότητα των δημόσιων ε, εισαγγελιών, τη διασύνδεση μεταξύ διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος, θέμα που αφορά ειδικότερα, ιδιαίτερα ορισμένες χώρες περισσότερο από άλλες. Όλες οι θεματικές παρουσιάσεις ανέφεραν ε, τον ε, ζήτημα του μηχανισμού παρακολούθησης είτε σε ευρωπαϊκό είτε σε εθνικό επίπεδο. Και πράγματι στη δική μας έκθεση θέλουμε να εξετάσουμε συστάσεις που έχουν ήδη γίνει από αυτόν τον μηχανισμό παρακολούθησης, ε, ιδιαίτερα τον ΟΕΣΑ, την γρέκο και τη σύμβαση κατά της ε, των εθνών κατά τη διαφθορά. Εξετάζουμε ιδιαίτερω την αξιολόγηση, τις αξιολόγησεις που έχουν γίνει στο σε αυτό το πλαίσιο και η πρόθεση μα βεβαίω είναι να μην υπάρξει επικάλυψη με στους του μηχανισμούς. Θέλουμε δεν θέλουμε να επαναλάβουμε τις εξαλλογήσεις που έχουν ήδη γίνει από αυτά τα όργανα, αλλά εκεί που οι συστάσεις δεν έχουν επαρκώς εφαρμοστεί ή υλοποιηθεί, θα θέλαμε να το επισημάνουμε και επίσης να χρησιμοποιήσουμε την έκθεση αυτή κατά της διαφθοράς ως μοχλό πίεσης για την καλύτερη εφαρμογή όλων αυτών των συστάσεων. Επίσης η διαφθορά στο ιδιωτικό τομέα βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής μας. Είναι τμήμα του πακέτου ε, κατά της διαφθοράς, εγκρίθηκε πέρσι από την Κομισιόν και επίσης έχουμε εγκρίνει το, τη δεύτερη έκθεση για την απόφαση πλαίσιο για τη διαφθορά στον ιδιωτικό τομέα που δεν δείχνει τόσο ικανοποιητικά αποτελέσματα όσον αφορά τη μεταφορά της ε, απόφασης ε, πλαίσιο. Ε, και για παράδειγμα την ε, ευθύνη των νομικών ε, προσώπων. Αυτό είναι ένας από τους τομείς όπου θα μπορούσαν να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα στο επίπεδο των χωρών μελών. Και σα ανέφερα προηγουμένω ότι η πρόθεση τη επιτροπή με την έκθεση αυτή είναι να επικεντρώσει σε ζητήματα εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο και στο νομικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό διεθνές επίπεδο. Και τέλος, θα ήθελα να, ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω πάλι για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσω εδώ και θα ήθελα να εκφράσω το ανοιχτό πνεύμα και τη διάθεση της Επιτροπής να σας συνδράμει με οποιοδήποτε τρόπο θεωρείτε ότι είναι δεδειγμένο συνεργαζόμενοι με την Επιτροπή ΚΡΙΜ ή στη συνέχεια όλων αυτών των θεματικών ομιλών πράγματα είναι ιδιαίτερως ε, χρήσιμα για μας ή σε σχέσεις σε σχέση με τις ε, ε, στατιστικές και τις συστάσεις που έχουν ήδη γίνει. Ε, θα συνεχίσουμε, εκ του θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγι σε αυτά τα θέματα. Ευχαριστούμε κυρία Στέφενοκ για τις διευκρινήσεις ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέλος ε, της συνθήκης του ΩΣΑ και το ΙΕ κατά της διαφθοράς. Είμαστε πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκή Ένωση στη συνθήκη του ΟΗΕ κατά της διαφθοράς, όχι στην αντίστοιχη συνθήκη του ΩΣΑ. Μάλιστα, ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Δεν ξέρω, πριν ολοκληρώσουμε, θα δώσουμε το λόγο για τη δευτερολογία στους συγκητές. Μπορεί να έχουν και άλλες ερωτήσεις να υποβάλουν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε πέντε λεπτά ο καθένας για τη δευτερολογία. Να δώσετε ερωτήσεις, να κάνετε κάποια σχόλια. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Γκαμπρίελ, ακολουθώντας την ίδια σειρά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι συνοπτική και επιγραμματική στις γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κάλυψε σε μεγάλο βαθμό, απαντώντας στον κύριο Νιούτον Ντάν για το πώς θα λειτουργήσει αυτό το σύστημα των κόκκινων σημαίων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει κάποια συγκεκριμένα μέτρα από το 2011 προκειμένου να δει πώς λειτουργεί ο μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της διαφθοράς και θέλουμε κάποια μέτρα που θα μας οδηγούν σε κοινούς δείκτες ε, και θέλουμε κάποιους δείκτες για να μπορούμε να εντοπίζουμε τη διαφθορά. Θα ε, θα κοινοποιείται ψηλό κόστο για συγκεκριμένα σχέδια, ζημιέ για τον προπολογισμό. Και επίση σε κάποιου ε, ανοιχτού διαγωνισμού θα πρέπει να δίνονται κάποιοι δείκτε ώστε να είναι κοινοί δείκτε και ένα σύστημα συναγερμού, προειδοποίηση. Δεν είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό που επινόησε το σύστημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε τι σχετικέ προτάσει και εγώ στο θεματικό μου έγγραφο ε, ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυ στην εξέλιξη του συστήματος αυτού ώστε να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα για το 2013, γιατί είχε προβλεφθεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι το, τα τέλη του 2012. Αλλά ίσως και το 2013 θα συνεχίσουμε ως Επιτροπή να ασχολούμαστε με το θέμα αυτό. Και επίσης, με βάση τις πληροφορίες που θα λάβουμε από τα κράτη-μέλη, θα μπορέσουμε και εμείς ως Επιτροπή να συμβάλλουμε με πολύ θετικό τρόπο στην παρακολούθηση του συστήματος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα σχόλια και τις παρεμβάσεις τους. Συμφωνώ με την πλειοψηφία των ε, σχολείων γιατί προσδιορίζονται οι προκλήσεις και τα διακυβεύματα του έργου της δικής μας Επιτροπής. Η κυρία Βερονίκ Ματιέ, η συντονίστρια του ΕΛΚ, επέμεινε στην ανάγκη τα κράτη-μέλη να ενσωματώσουν στην εθνική του νομοθεσία τουλάχιστον τι υπάρχουσε οδηγίε. Δηλαδή να ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε τι υφιστάμενε οδηγίε πριν αρχίσουμε να υποβάλλουμε νέες προτάσεις. Επίσης ευχαριστώ και την κυρία Φαγιόν γιατί επισήμανε την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Πώς θα μεταβιβάζονται τα δεδομένα, πώς θα συνεργάζονται καλύτερα τα κράτη-μέλη για να καταλήγουν σε κοινή δράση πανευρωπαϊκού χαρακτήρα. Επίσης, κάτι άλλο που ανέφερα στο εγγραφό μου είναι η επιτήρηση της εφαρμογής των συστάσεων της Όλαφ ή άλλων θεσμικών οργάνων. Γιατί πολύ συχνά εκεί προσκρούμε. Ποιες αρμοδιότητες έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποιες αρμοδιότητες έχει το ΔΕΚ και ποιες θα ήταν οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Αγγελικής Αρχής ενδεχομένω. Συμφωνώ πάντως με τους συναδέλφους, συμφωνώ με τα σχολεία τους και τους ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Κυρία... Γαμπριέλ ολοκλήρωσε. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Βάιλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πριν λοιπόν αναφερθώ στα δύο ερωτήματα που μου απευθύνατε, θα ήθελα να παραπέμψω τη γραμματεία σε ένα έγγραφο της Επιστημονικής Υπηρεσίας του Κοινοβουλίου για το θέμα της διαφθοράς για θέματα διαφθοράς και συμπεγνίας. Επειδή λοιπόν συζητάμε για την ε, σχετική οδηγία, νομίζω ότι όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα και ε, σε μία σελίδα αναφέρεται με λίγα λόγια πώς μπορούμε να αποφύγουμε την ε, διαφθορά και πού ακριβώς ελοχεύει ο κίνδυνος της διαφθοράς. Αυτή λοιπόν είναι μία μελέτη του Κοινοβουλίου ε, που την ανέθεσε σε μια Νορβηγίδα επιστήμων ε, και είμαστε και δύο στην Επιτροπή Κοινή Αγορά και ξέρετε γιατί το, θέτω, το, το θίγω το θέμα αυτό. Τώρα, όσον αφορά τι δύο ερωτήσει, δεν κατάλαβα καλά. Είπατε, κύριε Νιούτον Ντάν, πού διοχετεύονται τα χρήματα. Κοιτάξτε, υποθέτω, όχι μόνο στην Ιταλία. Τα χρήματα καταλήγουν όχι μόνο στην Ιταλία, αλλά και στους λογαριασμούς ε, των εγκληματιών. Ο κύριος Ταβάρες με ρώτησε κάτι άλλο. Ρώτησε ε, μήπως υπάρχουν ενδείξεις ότι ε, χρήματα από διαφθορά καταλήγουν στην πολιτική. Εγώ είμαι πεπισμένη ότι κυρίως στον τομέα της ε, δωροδοκίας κονδύλια αναμφίβολα καταλήγουν ε, σε πολιτικούς ε, σε όλα τα επίπεδα τοπική αυτοδιοίκηση σίγουρα και ανώτατο επίπεδο. Στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμών ε, εξετάζουμε μια τέτοια υποψία που υπάρχει. Αλλά κατά την άποψή μου αυτό δεν είναι οργανωμένο έγκλημα. Αυτά είναι ε, πολύ μεμονωμένες περιπτώσεις προσωπικού πλουτισμού και ιδιοτέλειας Γίνεται μία έρευνα για τη διαφθορά, ε, θα πρέπει να γίνει μία έρευνα για τη διαφθορά ε, από πολιτικά κόμματα ή σε πολιτικά κόμματα. Δεν ξέρω ε, τι συμβαίνει ακριβώ, αλλά σχετίζεται με τη διαφθορά. Και κοιτάξτε, η διαφθορά δεν αφορά μόνο την Ιταλία, αλλά πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε. Μιλάμε για τη δωροδοκία ε, και δωροληψία από πλευρά πολιτικών. Όλοι το γνωρίζετε αυτό. Αν δεν το έχετε ζήσει στο πετσί σας, το έχετε ακούσει. Άρα δηλαδή είναι σαφές ότι υπάρχουν όλα αυτά και πρέπει να προστατευτούν και οι δύο πλευρές. Δηλαδή τόσο το κράτος και την κοινωνία όσο και τους ε, πολιτικούς. Και οποτεδήποτε συμβαίνει κάτι ε, θα πρέπει να βγαίνει προς τα έξω και να τιμωρείται. Και υπάρχουν και δύο άλλα θέματα όπου ε, θέλω να τα διευκρινίσουν ε, οι πρώτη Επιτροπής και η Γραμματεία. Είπατε ότι μεταφράζονται τα θέματα που παρουσιάστηκαν άκουσα ότι δεν μεταφράζονται. Αν τελικά μεταφραστούν αυτό θα ήταν πάρα πολύ καλό γιατί εγώ θα μπορούσα με όλα τα θέματα που συζητήσαμε σήμερα εδώ να κάνω πολλή δουλειά στη Γερμανία να ευαισθητοποιήσω τους πολίτες ε, να μεταφέρω πολιτικές πληροφορίες εφόσον βέβαια μεταφραστούν οι ομιλίες. Και κυρία Γκάμπριελ δεν ξέρω ίσως ε, η γραμματεία της Επιτροπής να έρθει σε επαφή με τη γραμματεία της ε, ΙΜΚΟ. Ε, θα ψηφίσουμε σύντομα για την έκθεση Ταραντέλα για τον εξυγχρονισμό ε, των δημόσιων συμβάσεων. Και αν τελικά προκύψει ότι πρέπει να συμπεριλάβουμε ένα συγκεκριμένο εντάφιο με το οποίο να συμφωνούμε όλοι μας ε, ότι δηλαδή θα πρέπει να αναφέρουμε και μέτρα πάταξης της φοροδιαφυγής αυτό ε, θα ήταν ε, πάρα πολύ επικοδομητικό. Τελευταία παρατήρηση για να σας καθησυχάσω. Το αργότερο, το φθινόπωρο του επόμενου έτους, η Γερμανία μετά από την αλλαγή πολιτικής που θα υπάρξει σε εμά θα υπογράψει και την οδηγία περί διαφθοράς. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ σε ό,τι φορά τη μετάφραση των θεματικών εγγράφων. Ε, το έγγραφο εργασία του κυρίου Κολίνου είναι αυτό που θα μεταφραστεί, όχι τα θεματικά έγγραφα. Το περιεχόμενο των θεματικών εγγράφων ε, θα συμπεριληφθεί στο έγγραφο εργασία του κυρίου Γιακολίνου. Αυτό έγινε και αυτό βρίσκεται σε διαδικασία μετάφραση. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν εδώ συνεργάτε του κυρίου Γιακολίνου, τα σημειώνουν κατά λεπτό όλα αυτά. Και πολλά από τα στοιχεία των θεματικών εγγράφων θα συμπεριληφθούν στο έγγραφο εργασία του κυρίου Γιακολίνου. Κυρία Βάιλερ. Παρόλο που δεν το προσδιορίσα, όταν σα έκανα την ερώτηση, είχα κατά νου το θέμα των ευρωπαϊκών ταμείων που χρηματοδότησαν επιχειρήσεις, το, οι οποίες στη συνέχεια νόμιμα συμμετείχαν ε, σε κομματική χρηματοδότηση. Μπορεί να μην μου σαφή την ερώτησή με αυτό εννοούσα πάντως προηγουμένως. Ναι, ε, ξέρω τι εννοείται και δεν θεωρώ ότι αποκλείεται εντελώς, παρόλο που δεν μπορώ να το φανταστώ. Αλλά στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ρωτήσουμε την Όλαφ ή έστω και την Κομισιόν αν ε, έχει τέτοιες ενδείξεις. Άκουσα κάτι για τη Σερβία, αλλά εκεί δεν πρόκειτο για ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά για μία κονδύλια από ευρωπαϊκά ταμεία, αλλά άλλες πηγές. Αλλά τελικά ε, μπόρεσαν να το αναστείλουν με, χρησιμοποιώντας ένομα μέσα και επιβολή κυρώσεων, ποινικών κυρώσεων. Ε, εν πάση περιπτώσει όλα είναι δυνατά στον κόσμο μα, αλλά εγώ δεν ξέρω καμία τέτοια συγκεκριμένα περίπτωση. Ευχαριστούμε κυρία Βάιλερ. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Σκυλακάκη. Ευχαριστώ. Όλοι ε, έχουμε υπόψη τέτοιε υποθέσει αυτή που αναφέρατε στην τελευταία σα ερώτηση, τουλάχιστον στη δική μου πατρίδα αλλά και σε άλλες φαντάζομαι ευρωπαϊκές χώρες. Είχαμε υποθέσεις, τεράστιες, ε, πολύ σημαντικές υποθέσεις δωροδοκιών που ερευνώνται για χρηματοδότηση κομμάτων και μάλιστα μερικά από τα κονδύλια αυτά προέρχονταν από ευρωπαϊκά ταμεία. χωρίς μικρόφωνο δυστυχώς το σχόλιο της κυρίας Βάιλ. Και η ζήμες εξαίρεση είναι αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς ε, χωρίς μικρόφωνο γίνονται τα σχόλια από την αίθουσα. Είχαμε πολύ σημαντικές υποθέσεις και επανέρχομαι στην ουσία του εγγράφου μου. Θα ήθελα πρώτα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν μπορεί να κάνει πιο λεπτομεριακά σχόλια και παρατηρήσει για τα θεματικά έγγραφα. Νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ και τον εισηγητή μας, τον κύριο Γιακολίνο, να έχουμε μια πιο διεξοδική ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα αυτό. Τα θέματα δηλαδή που πραγματεύονται τα έγγραφά μας. Δεν είχα προηγουμένως την ευκαιρία να αναφερθώ σε Συγκεκριμένε συστάσει προηγουμένω. Θα ήθελα τώρα να το κάνω, αν μου επιτρέπετε, δεν θα με ακρηγορήσω Πέραν τη γενική αρχή ότι χρειαζόμαστε πιο ισχυρά θεσμικά όργανα και φορεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση, την πάταξη της διαφθοράς, ώστε να μπορέσουμε και εμείς όπως οι Αμερικανοί να έχουμε αποτελεσματική πολιτική κατά της διαφθοράς, πέραν αυτής της ε, ανάγκης, πιστεύω ότι χρειαζόμαστε και ένα πανευρωπαϊκό αποτελεσματικό σύστημα προστασίας των ε, whistleblowers, των καταγγελόντων, των πληροφοριοδοτών, γιατί υπάρχουν ε, χώρες, έχουμε ορισμένε χώρες όπου αν κάποιος καταγγέλων ε, εμφανιστεί στις αρχές της δημόσιας αρχής δεν ξέρω τι θα του συμβεί στο, στο τέλος. Μένει τελείως απροστάτευτος και δεν υπάρχει ούτε πανευρωπαϊκή προστασία. Η μόνη προστασία που μπορεί να περιμένει είναι από τις εθνικές αρχές και πολύ συχνά οι εθνικές αρχές δεν έχουν αποτελεσματικά συστήματα προστασίας των καταγγελόντων. Μόνο δύο από τις 27 χώρες μας λέει η διεθνή Διαφάνεια ότι έχουν αποτελεσματικά συστήματα προστασίας των ανθρώπων, αυτών που κάνουν καταγγελίες και δίνουν πληροφορίες για περιστατικά διαφθοράς. Επίσης πρέπει να έχουμε ένα κατάλληλο ποσοστό, 50% των ε, ερευνών με πρωτοβουλία της ΟΛΑΦΑ να ερευνώνται. Γιατί αυτή τη στιγμή ε, ερευνούμε μόνο πληροφορίες που μας δίνονται. Δηλαδή, αν έχουμε ένα κύκλωμα οργανωμένου εγκλήματος και ε, διαπράττεται εγκλήματα κανένας δεν πρόκειται να σας ελέγξει. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε με τα, με τα κοινοτικά κονδύλια στον τομέα σας στη χώρα. Χρειαζόμαστε και αυτεπάγγελτες έρευνες ίδιας πρωτοβουλίας. Τουλάχιστον το 50% να είναι αυτεπάγγελτες έρευνε. Να μην ε, επιλαμβανόμαστε μια υπόθεση, μια έρευνα μόνο μετά από καταγγελία. Να υπάρχει δυνατότητα και με ίδια πρωτοβουλία αυτεπάγγελτα να ε, ξεκινούμε Επίση, Επίσης, ε, να μπορούμε να κάνουμε άμεση συγκρίσεις ε, των τιμών αγαθών και υπηρεσιών. Αυτό θα ήταν πολύ ενδιαφέρον ε, για τις ε, δημόσιες προμήθειες και την πάταξη της διαφθοράς εκεί. Γιατί αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ των τιμών των προσφορών και μπορεί ε, και να μην γνωρίζει κανείς τη διαφορά, ούτε καν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορεί κανείς να αγοράζει το ίδιο πράγμα δεκαπλάσια, δεκαπλάσια τιμή και κανείς να μην ανακαλύψει αυτή τη τεράστια διαφορά των τιμών. Επίσης, θεωρώ ότι θα πρέπει να προωθήσουμε την έρευνα της χρήσης των νέων τεχνολογιών και των διαφορών συστημάτων ελέγχου και να διευκολύνουμε την εφαρμογή τους. Για παράδειγμα, έλεγχη στους φόρους, φορολογική έλεγχη. Γιατί να μην μπορούμε να κάνουμε online, ε, να, να δίνονται online πληροφορίες για το φορολογικό έλεγχο, τη στιγμή δηλαδή που πραγματοποιείται από την εφορία ασκείται έλεγχος φορολογικός σε μία επιχείρηση, γιατί να μην γίνεται αυτός ε, online, απευθείας να μεταδίδεται, ώστε να μπορούν οι προϊστάμενοι να, ή οι αρμόδιες για τη, κατά της διαφθοράς αρχές να ελέγχουν την κατάσταση. Γιατί αυτή τη στιγμή όλοι οι έλεγχοι ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα σε κράτη-μέλη που υπάρχει έντονο το φαινόμενο της διαφθοράς, γίνονται με διαφανή τρόπο. Θα πρέπει αυτή την αδιαφάνεια να την καταπολεπίσουμε, γιατί σε πολλά ε, σε πολλές περιπτώσεις είναι συστημική διαφορά, ε, η διαφθορά, χρόνια διαφθορά, ενδημική. Επίσης, ε, να αυξήσουμε του σπόρους των φορέων που ασχολούνται με την προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και ένα σημαντικό τμήμα του προϋπολογισμού τους να το συνδυάσουμε με τις επιδόσεις τους ό,τι αφορά την διαχείριση των κονδυλίων. Γιατί αυτή, σήμερα όχι μόνο δεν έχουμε αρκετούς σπόρους, αλλά συνεχίζουμε τις περικοπές. Να πούμε λοιπόν στους αρμόδιους φορείς. Θα σας δώσουμε θα, επιβραβεύσουμε τις επιτυχίες σας ε, ενισχύοντας τους πόρους για να αυξήσετε και εσείς τις ερευνές σας. Γιατί χωρίς έρευνες και χωρίς εξυχνίαση των περιπτώσεων αυτών πώς θα είμαστε αποτελεσματικοί. Ευχαριστούμε κύριε Σκυλακάκη η, χώρα για την οποία ακούμε όλο και περισσότερες ε, πληροφορίες ε, για παράνομη χρηματοδότηση των κομμάτων από κοινοτικά κονδύλια δεν είναι η Ελλάδα, είναι άλλη χώρα που είχα στο μυαλό. Για άλλη χώρα ακούμε πληροφορίες, ο κ. Δε Ε, καταρχήν θα ήθελα να έρθω στα σχόλια της κυρίας Ματιώ όσον αφορά την ε, μεταφορά των νομικών διατάξεων. Όσον αφορά την ενιαία αγορά έχουμε την έκθεση ΣΟΑΠ που ασχολείται με το θέμα της διακυβέρνησης της αγοράς και την ε, προσπάθεια να υπάρξει ένα σύστημα το οποίο να είναι πιο δεσμευτικό ε, ε, μέσα στο οποίο να μπορούν να υπάρξει μια καλύτερα εφαρμογή. Επίσης, διαδικασίες επί τη παραβάση σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θα παρουσιαστούν σύντομα τα σχετικά αποτελέσματα στο Κοινοβούλιο. Το πρόβλημα είναι ότι η διαφθορά ποτέ δεν έχει αναγνωριστεί ως τμήμα της ενιαίας αγοράς. Η Σύμβαση δεν το θεωρεί επισήμως ως τμήμα του κοινοτικού κεκτημένου. Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο, θα έπρεπε να προσαγγιστεί στο επίπεδο αυτό σε σχέση και με τον θεμητό ανταγωνισμό και με τον τρόπο αυτό θα πρέπει να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση προς τις χώρες μέλη για να εφαρμόσουν τη σύμβαση με τον ΩΣΑ αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει και ίσως θα πρέπει να αναφερθεί αυτό πιο ρητά στην έκθεση. Τώρα, όσον αφορά τα όσα είπε ο κ. Νιούτον Ντάν, ε, τι να πω ε, σε σχέση με τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου. Απλώς θα μπορούσα να πω ότι το κόμμα το οποίο εκπροσωπώ εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι πολύ υπέρ της εκχώρησης ε, κυριαρχίας και εθνικών αρμοδιοτήτων και ένας ε, τομέας όπου είναι αναγκαία η σωστή συνεργασία ε, είναι η προσπάθεια πάταξης του οργανωμένου εγκλήματος γιατί βεβαίως οι εγκληματίες δεν ε, σέβονται τα εθνικά σύνορα και αν κάποιος άδικο πραγεί στην Ιρλανδία θα πάει και στην, και στη Μεγάλη Βρετανία θα πάει και στη Μεγάλη Βρετανία. Ε, ε, οι άλλες μου παρατηρήσεις αφορούν ε, την Κομισιόν. Καταρχήν θα πρέπει να πω ότι υπάρχουν κάποιες αναφορές στις προτάσεις για τις δημόσιες προμήθειες που αναφέρονται στο θέμα της σύγκρουσης ε, συμφερόντων. Εάν πάρουμε για παράδειγμα τις διατάξεις ε, για, την ε, για τη συμπερίληψη των εταιριών σε έναν κατάλογο που έχουν κάνει κάποιες παραβιάσεις για, στον τομέα των δημοσίων προμηθειών, μια τέτοια μαύρη λίστα. Νομίζω ότι πράγματι έχετε αποβάλει πολύ θετικέ ε, προτάσει στην Κομισιόν στην κατεύθυνση αυτή και θεωρώ ότι ίσω είναι καλή. Ε, ε, δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα να επανέλθει ένα χρόνο μετά. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε με την υποβολή μιας έκθεσης μέχρι πάρουμε από εσά τις εκθάσεις για την νομοθεσία. Αναφέρθηκα στο θέμα της ευθύνης των νομικών προσώπων επί παραδείγματι. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ βασικό για οποιαδήποτε προσπάθεια στον ε, ποινικό τομέα. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει σαφήνεια στον τομέα αυτό, καθώς και μια σαφήνεια ε, όσον αφορά την ευθύνη της κεντρικής εταιρεία ε, έναντι των θηγατρικών. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται με κάποιες ποινικέ προτάσεις, ε, με κάποιε προτάσει σχέση με το ποινικό νόμο ε, χωρί να συμπεριλαμβάνεται όλα αυτά τα θέματα, δηλαδή μια οριζόντια προσέγγιση. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε περισσότερε προτάσει για να έχουμε αυτή την οριζόντια προσέγγιση. Ε, θέματα για παράδειγμα πως είναι οι διευκολύνσεις, οι οικονομικές διευκολύνσεις ή το θέμα των καταγγελώντων, των whistleblowers που ανέφερε ο κύριος Σκυλακάκης. Τέλος, αναφέρατε, η Κομισιόν ανέφερε και πάλι το θέμα ε, το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τμήμα, ε, έχει, συμμετάσχει, είναι μέλος μάλλον της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών. Και εγώ πολύ συχνά είμαι ιδιαίτερος απογοητευμένος για το θέμα ότι η Κομισιόν δεν είναι υπόλογη σε σχέση με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Εάν ζητούνται κάποια πράγματα από τις χώρες μέλη, νομίζω ότι είναι η Κομισιόν αυτή η οποία θα πρέπει να δίνει το καλό παράδειγμα και να υποβάλει κάποιες αναφορές. Η Κομισιόν θέλει να έχει ακριβώς το καθεστώς του παρατηρητή για να αποφεύγει να υπεκφεύγει τις υποχρέωσεις του να ε, υποβάλει κάποιες αναφορές, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι σωστό αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Νταλουκάς ε, δεν ξέρω εάν θέλει να πάρει τον λόγο για μερικά λεπτά για να απαντήσει στις ερωτήσεις που έγινε επιτέλους από τον κύριο Ντε Γιόγκ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, καταρχήν, ε, πραγματικά θα δώσουμε κάποια γραπτά σχόλια για τις θεματικές ε, ομιλίες. Και σε σχέση με το είπε πράγματι έχουμε αυτή την υποχρέωση ε, επειδή είμαστε πλήρες μέλος, να συμμετάσχουμε και στο μηχανισμό παρακολούθησης που λειτουργεί από το 2009. Θα ήθελα απλώ να υπογραμμίσω ότι, να υπογραμμίσω δεν είναι μόνο η Κομισιόν η οποία είναι υπόλογη όσον αφορά την υποβολή αυτών των αναφορών, αλλά ε, είναι υποχρεωμένα να το πράξουν και όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υπάρχουν παρόμοια θέματα τα οποία έχουν τεθεί και στην Γκρέκο ε, και υπάρχουν κάποιοι λόγοι για το ότι δεν ε, έχει γίνει μέχρι στιγμής αυτή η υποβολή αναφορών, γιατί θα πρέπει να διευκρινιστούν προηγουμένως κάποια συγκεκριμένα νομικά θέματα τα οποία αφορούν αυτή την αναφορά εκ μέρους των θεσμικών οργάνων. Άρα δεν πρόκειται για ένα θέμα λοιπούς βούλησης και συμφωνώ μαζί σας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δώσει το καλό παράδειγμα στο πλαίσιο αυτό της συνεργασίας με τα Ηνωμένα Έθνη ή σε σχέση με τη συμμετοχή της στην ε, Γκρέκο και ήταν μία από τις τελευταίες προτάσεις που έκανε ο πρόεδρος κ. Μπαρόζο για τη συμμετοχή στην Γκρέκο και θα πρέπει επίσης να προβαίνει σε κάποιες ε, ε, διευκρινήσεις συγκεκριμένων νομικών πτυχών για την αξιολόγηση των θεσμικών οργάνων στη βάση των συνθήκων. Ε, δεν αφορά λοιπόν αυτό το ζήτημα μόνο την Κομισιόν, αλλά τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το θέμα της υποβολής αναφορών. Τώρα, όσον αφορά την προστασία των whistleblowers, πράγματι έχουμε την επίγνωση ότι αυτό είναι ένας μέσο όπου οι χώρες μέλη δεν ε, έχουν μέχρι στιγμής επαρκή ε, προστασία αυτού και του δημόσιο για τον ιδιωτικό τομέα. Γι' αυτό η Κομισιόν αυτή τη στιγμή διεξάγει μια έρευνα για να έχει μια εποπτεία όλων των, ε, του συνόλου της νομοθεσίας των χωρών μελών σε σχέση με τους whistleblowers για να δούμε ποια πολιτική θα πρέπει να χαράξουμε στο τομέα αυτό. Όσον αφορά το blacklisting των επιχειρήσεων, των εταιριών, ε, πράγματι το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερο καυτό και συμφωνώ μαζί σα ότι σε ορισμένε περιπτώσει θα μπορεί να είναι ιδιαίτερο χρήσιμο εργαλείο για την πάταξη διαφθορά. Αλλά επίσης δεν πάβει να είναι ένα θέμα το οποίο γύρει κάποια θέματα, για παράδειγμα σχέση με την προστασία δεδομένων. Και από τις χώρε μέλη είναι πολύ λίγα αυτά τα μέλη που δημοσιοποιούν ε, τα, τις, ε, τους καταλόγους ε, για τις υποβολές ε, προσφορών για τις δημόσιες προμήθειων. Ε, δημόσιων, για προμήθειες, συγγνώμη. Ε, και ε, ε, θεωρώ ότι το σημείο αυτό είναι ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και όταν κάνουμε την αξιολόγηση της έκθεσης για την πάταξη διαφοράς θα συμπεριλάβουμε αυτό το θέμα. Ένα τμήμα αυτής της έκθεσης Βεβαίω ε, θα περιλαμβάνει κάποιες ε, συγκεκριμένες συστάσεις, αλλά και συστάσεις για μελλοντικέ δράσει τη Ευρωπαϊκής Ένωσης νομοθετική ε, φύσεως. Και βεβαίω αυτό θα εξαρτηθεί από τα συγκεκριμένα ευρήματα που θα έχουμε στο πλαίσιο των εξολογήσεων. Σας ευχαριστώ. So, thank Και εμείς σας ευχαριστούμε κυρία Στεφανούκ. Υπάρχουν και συστάσεις ε, προς εμάς. Πριν λοιπόν ε, κλείσουμε την ε, συζήτηση, θα ήθελα ε, να διαβάσω την πολύ συγκεκριμένη σύσταση του κ. Ντεγιόγκ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συγκεντρώνει πληροφορίες. Ε, επίσης υπάρχουν οι συστάσεις στο οσα που θα πρέπει να συζητηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο θα πρέπει να καταθέσει στάσεις για το σύνολο της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αναφέρεται και ο μηχανισμός Γκρέκο. Πρόκειται λοιπόν ε, για την εφαρμογή αυτών των συστάσεων. Αν δεν υπάρχει τίποτα άλλο και δεν νομίζω ότι υπάρχει, κλείνουμε τη συνεδρίασή μας. 23 ε, Ιανουαρίου είναι η επόμενη συνάντηση από τις 9.30 και από τις 3 ε, μέχρι τις 6.30 και 24 Ιανουαρίου το πρωί. Γεια σας.